So, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και σας ευχαριστώ ε, ιδιαίτερα για τα περαστικά που μου στείλατε για την ασθένειά μου. Οι συνάδελφοι εδώ πέρα δεν ξέρω τελείωσαν με τα τεχνικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα περαστικά που μου στείλατε. Θέλω να παρατηρήσω. Εντάξει, 7-8 μήνες δεν είναι απλή υπόθεση και όταν έχει κάποιος μία σχέση κάπως με τα βρυξελιώτικα αντιλαμβάνουμε πόσο δύσκολο είναι να παρακολουθήσει κανείς ένας πολίτης το τι κάνουμε εμείς εδώ. Το πώς ε, θα τελειώσουν τα πράγματα δεν ξέρω, αλλά είναι σαν να κοιτάει κανείς με τα κιάλια προς τις Βρυξέλλες, δεν βλέπει όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι όπως είπα. Περνάμε στην μερίσια διάταξη λοιπόν. Σημείο 11, το 11 πρέπει να αναβληθεί. Θα πάει στις 28 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τις γλώσσες τις έχουμε όλες πλην ε, της ε, Κροατικής ε, και Ιρλανδικής ε, και τα Μαλτέζικα θα τα χάσουμε για μία ώρα, αλλά ο Ντέβιτ Κάζα δεν θα είναι εδώ, οπότε δεν υπάρχει και θέμα. Μετά έχουμε μία αλλαγή της σύνθεσής μας. Η ε, ε, Άννε Σέντερ, αν βλέπω καλά, θα αντικαταστήσει εδώ την κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ και μας έχει εγκαταλείψει η κυρία Μισελ Αλιό από την θέση της ως αναπληρωματικό μέλος. Δεν μου έχουν πει ποιος θα την διαδεχτεί. Λοιπόν, και έχουμε και κάποια ευχάριστα. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από τον τέταρτο τριμερή διάλογο για τις ε, καρκινογόνες ε, και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Ε, τις λεπτομερίες δεν τις γνωρίζω ακόμα. Θα ψηφιστεί 30 Αυγούστου στην Επιτροπή μας. Από ό,τι φαίνεται πήγαν καλά τα πράγματα για τις θέσεις μας το θέμα αφορά 100.000 άτομα τα επόμενα 50 χρόνια που θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τον καρκίνο αυτό σε μια πρώτη φάση να ευχαριστήσω λοιπόν εδώ πέρα την Μαρίτα που έκανε πολύ καλή διαπραγμάτευση και να την ευχαριστήσω και προσωπικά τη Μαρίτα και όλους τους αντιπροέδρους για την στήριξή τους ε, κατά την απουσία μου. Ε, με αντικαθέστησα νομίζω επάξια, με κάποιες συγκρούσεις από την άποψη, αλλά νομίζω όλα καλά πήγανε. Είχαμε και μία αντιπροσωπεία για το Ταλίν υπό την ηγεσία του Καλβεν Έχουμε και τη σχετική έκθεση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα, δεν υπάρχει χρόνο σήμερα. Και τελευταίο, έχουμε τα πρακτικά της 21 η 22ης Ιουνίου και 29 η 30ης Μαΐου. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Όχι, οπότε περνάμε στο σημείο 4 ο αντίκτυπος των επιχειρηματικών μοντέλων συμπεριλαμβανομένης της συνεργατικής οικονομίας, στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας απασχολήσει ε, αυτό το θέμα σήμερα, εδώ και κάτι μήνες ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Έχουμε και μια σημαντική συνεισφορά για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε 15 Ιουνίου. Σήμερα θέλουμε να εμβαθύνουμε υπό μορφή ακρόασης και καλωσορίζω τέσσερις ειδικού. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Μπεντουέ, Senior Marketing Consultant ε, Social Economy Island, τον Ρόναλντ Ιούντικ, Γενικό Γραμματέα της Uni Europe, ε, του Συνδικάτου των Υπηρεσιών Στίβ Μπέρκε, ο οποίος είναι οικονομολόγος του ΩΣΑ και τον καθηγητή Μάρτιν Ρίσακ του Πανεπιστημίου της Βιέννης, καθηγητή εργατικού δικαίου. Περνάμε λοιπόν αμέσως ε, στις παρουσιάσεις σας. Σας παρακαλώ να περιοριστούτε σε 10 λεπτά. 10 ε, λεπτά ο καθένας, ε. Έχετε χρόνο. νομίζω φτάνει ο χρόνος και αν δεν ξεπεράσετε θα σας το πω εγώ. Λοιπόν, κυρία Ντουέ, έχετε τον λόγο. Οι κυρίες προηγούνται. Microphone, please. Sorry, yes, sorry about that. So thank you, Chairman, and good morning to all members, distinguished guests, ladies and gentlemen. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ε, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε για αυτήν την ε, δημόσια ακρόαση. Είναι για μια ευκαιρία η οποία προέκυψε από μια συζήτηση που είχα με έναν Ιρλανδό Ευρωβουλευτή σε μια συνάντηση στο Σκιβερίν στην Κομιτεία του Κόρκ και αφορούσε ακριβώς την πάρα πολύ γρήγορη σύνδεση του διαδικτύου σε ένα κτίριο στην περιοχή αυτή που έκανε ένα παλιό κτίριο κινηματογράφου σε, ε, το μετέτρεψε σε ένα έργο και ένα χώρο συνεργατικής ψηφιακής οικονομίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον βουλευτή για την πρόσκληση. Λοιπόν, είμαι ιδρυτικό μέλος της Sharing Economy Ireland, ε, μια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί διάφορα ε, μέρη από διεθνείς εταιρείες μέχρι Ιρλανδικές ε, νεόφυης επιχειρήσεις. Και έχουμε, εκπροσωπούμε Διαφορετικέ φωνές και εμπειρία. Και τα ερωτήματα είναι πώ εργάζονται οι εργαζόμενοι του 21ου αιώνα και τι μορφή θα πρέπει να έχει το δίκτυ ασφαλείας του 21ου αιώνα. Μια περίπλοκη συζήτηση που βασίζεται σε συγκεκριμένη έρευνα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια επίσης συμμετείχα σε έρευνα για τη συνεργατική οικονομία στην Ευρώπη και έτσι κατάφερα να έρθω σε επικοινωνία με ιδρυτές επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και με μικροεπιχειρηματίες που ξεκινούν τώρα. Επίσης ήρθα σε επαφή με τα άτομα τα οποία προωθούν και φιλοξενούν επιχειρήσεις της συνεργατικής οικονομίας. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τα ζητήματα που απασχολούν την Επιτροπή σας. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθώ στην δική μου εμπειρία, την εμπειρία της συνεργατικής οικονομίας, την Ιρλανδία για τα ζητήματα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης στον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα θα πω ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια του πώς αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα την οικονομία και το τι σημαίνει αυτό για την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να δούμε και τις συνεισφορές και τις προκλήσεις αυτών των αλλαγών και να συνεργαστούμε για να βρούμε κάποιες λύσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να δούμε τους διάφορους όρους. Σήμερα μιλάμε για μια οικονομία συνεργατική που λέγεται επίσης και οικονομία πλατφόρμας. Υπάρχει επίσης η γίγα οικονομία, η οικονομία των εφαρμογών και διάφοροι άλλοι όροι. Αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος όρος που είναι αποδεκτός από όλους. Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω τον όρο συνεργατική οικονομία και ε, οικονομία του διαμοιρασμού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν του Ιουνίου του 2016. Βεβαίω η ορολογία διαφέρει, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες πόλεις οι οποίες εντάσσονται στην συμμαχία των πόλεων που ξεκίνησε στο Άμστερνταμ. Η οικονομία αυτή αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ιρλανδία και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα Προκύπτει λοιπόν από πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τα κάτω για να προωθήσει την υπεύθυνη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας. Και βλέπουμε τα διάφορα μέλη της οικονομίας αυτής στην Ιρλανδία φέτος ε, κάποια στιγμή οι χρήστες και οι πάροχοι αυτών των πλατφορμών θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη τους. Και ακριβώς ε, θέλουμε να έχουμε μέλη από όλες τις πτυχές για να έχουμε μια όσο δυνατόν ευρύτερη συζήτηση. Έχουμε τέσσερα λοιπόν βασικά θέματα. Ευθύνη, εμπιστοσύνη, έξυπνη ρύθμιση, ευκαιρίες για την Ιρλανδία και πρακτικές εργασίας. Όπως είπαμε, η σαφήνεια θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να έχουμε καλύτερες συζητήσεις, να αντιληφθούμε καλύτερα το πόσο διαφορετικά είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα τον Δεκέμβριο 2016 η έκθεση του Κοινοβουλίου για την συνεργατική οικονομία λέει ότι η οικονομία αυτή δεν είναι μονολυθική, αλλά χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία επιχειρηματικών μοντέλων. Έτσι, δεν μπορούν να δημιουργηθούν ενιαία μέτρα, αλλά αυτό προσφέρει και ευκαιρίες για νέα είδη εργασίας. Συγγνώμη, ναι, η σαφήνεια επίσης για το μέγεθος έχει μεγάλη σημασία. Όταν έχουμε τις ίδιες διεθνείς πλατφόρμες οι οποίες κυριαρχούν στην συζήτηση, οι οποίες όμως δεν είναι ενδεικτικές για όλες τις πλατφόρμες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του ζητήματος, μόνο μια πολύ μικρή ομάδα πλατφορμών έχουν πάνω από 100.000 μοναδικούς ημερήσιους επισκέπτες. Οι περισσότερες πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επιχειρήσεις όπως το Rent My Dress, ε, μια μικροπλατφόρμα που επιτρέπει στις γυναίκες να νοικιάζουν τα ρούχα τους, ή το Τσάιλο, μια άλλη ερλαντική επιχείρηση που επιτρέψει ο κόσμος να νοικιάζει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, από μικρά τλεκατευθυνόμενα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Επίσης η το Τσάιλο, μια άλλη Ιρλανδική επιχείρηση που επιτρέπει στον κόσμο να νοικιάζει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανεί από μικρά τηλεκατευθυνόμενα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Επίσης, η σαφήνεια θα μας βοηθούσε στο να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται το όρος γίγα οικονομία, οικονομία των γιγαμπάιτ. Επίσης είναι αρκετά ενδεικτικός ε, όπως επίσης ε, και η οικονομία των εφαρμογών. Μια πρόσφατη μελέτη της McKinsey λέει ότι 20 30% του, εργα... του ενεργού πληθυσμού σε ήπα και Ευρώπη έχουν κάποια έπαφη με το αντικείμενο. Για το 96% των ανεξαρτήτων εργαζομένων οι επαφές είναι κυρίως offline και τα κοινωνικά ωφέλη και επιδόματα κατά κανόνα δεν σχετίζεται με το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι ασχολούμενοι στον τομέα αυτών βεβαίως θα το δέχονταν πολύ ευχάριστα. Το πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για μια Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Συνεργατική Οικονομία εστιάζει στι πολλές ευκαιρίες και ωφέλη που έχει αυτό ο κλάδος αλλά και τι προκλήσει που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ακριβώς αυτή την διπλή προσέγγιση, να συνεργαστούμε για να δούμε τις προκλήσεις χωρίς να ξεχνάμε το τι προσφέρουν αυτές οι καινοτομίε στον κόσμο, στην κοινωνία και στην ευρύτερη κοινότητα. Μία από αυτές είναι η ποικιλομορφία που προσφέρει πρόσβαση στην εργασία σε νέους, γυναίκες, ηλικιωμένους, ανάπηρους και παραδείγματα τα βλέπουμε σε πλατφόρμες όπως το Employee Mom, μια ελληνική πλατφόρμα που φέρνει τους γονείς σε επαφή με εταιρείε οι οποίες έχουν κάποιες εναλλακτικέ θέσεις εργασίας ή μια άλλη Ιρλανδική ε, startup ε, η οποία φροντίζει για ηλικιωμένα άτομα ή το έντεκο το οποίο ε, προσφέρει την δυνατότητα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες να βρουν προσβάσιμα ξενοδοχεία και διάφορα μέρη για να πάνε διακοπές. Μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη συμπερίληψη πολλών ατόμων, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό ε, χωρίς να υπάρχει κάποιος αποκλεισμός. Η συνεργασία μεταξύ πλατφορμών, κρατών, συνδικάτων, ασφαλιστών έχει μεγάλη σημασία για τον 21ο αιώνα για να βρούμε τις λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους εργαζόμενους του 21ου αιώνα. Επίσης, μπορούμε να δούμε το τι γίνεται με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά παρόλα αυτά να προσφέρουν λύσεις οι οποίες είναι ευέλικτες και αναλογικές, όπως παραδείγματι το Smart, μια συνεταιριστική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1998 και προσφέρει τώρα υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για να παρέχει ακριβώς παροχές σε διαφορούς εργαζόμενους. Ή το Dimly από την Δανία που επιτρέπει ακριβώς την πιστοποίηση της ε, ταυτότητας και της δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δοκιμών σε ένα περιβάλλον ε, στο διαδίκτυο υπό την αίρεση πάντα διαφόρων περιορισμών. Εν ολίγης, ε, υπάρχουν πολλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες στη συνεργατική οικονομία για άτομα, εταιρείες και κράτη, αλλά και προκλήσεις για τον κόσμο της εργασίας σε μια ψηφιακή οικονομία η συνεργατική οικονομία, το Sharing Economy Island, η οργάνωσή μα, στόχο είχε ακριβώ να προβλέψει τα κρίσιμα ζητήματα και να αναλάβει κάποιε υπεύθυνε πρωτοβουλίε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με το φόρουμ ε, της ε, Κομισιόν που θα γίνει τον Οκτώβριο στο Δουβλίνο και είχαμε λάβει μέρος ε, και σε ένα ανάλογο φόρουμ στην Λισαβόνα και στην Μάλτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω την περαιτέρω συζήτηση. Ich bin beeindruckt über die Εντυπωσιάστηκα από το πώς στηρίσατε και τον χρόνο. Εντυπωσιάστηκα με ακρίβεια δευτερολέπτου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο στον Ολίβιε Ρέτυχ να μας δώσει την άποψή του για το Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για την πρόσκληση αλλά και για την καλή συζήτηση που είχαμε πέρσι για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θα προσπαθήσω να τηρήσω και εγώ το χρόνο μου. Καταρχάς να πλαισιώσω λίγο τη συζήτηση και να αναφέρω κάποια στοιχεία που εμείς ως συνδικάτα θεωρούμε σημαντικά όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση. Για τη Union Europa η κυριότερη πρόκληση σήμερα είναι οι κανονισμοί, η κοινωνική ασφάλιση και η απασχόληση θα πρέπει να συνοδεύουν τα παρουσιακά μοντέλα του επιχειρήν. Και εδώ αυτή η μορφή οικονομία που συζητάμε είναι ένα παράδειγμα. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα κάποιε τάσει. Η πρώτη είναι το ότι οι επιχειρήσει ε, καλύπτουν όλο και μικρότερο κομμάτι στην ε, αλυσίδα αξία. Μετά διασυνοριακά παράγονται προϊόντα και υπηρεσίε που καλύπτουν καταναλωτέ και πελάτε. Και το τρίτο είναι ότι οι επιχειρήσει χρησιμοποιούν όλο και, όλο και λιγότερο εργατικό δυναμικό. Οπότε αυτό που θεωρούμε ως ιστροή πρέπει να συμπληρώνεται από αυτοαπασχολούμενους, από μη απασχολούμενου και από εξωτερικές συμβάσεις, από αναθέσεις και υπεργολαβίες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ με τους νομοθέτες και με τα συνδικάτα σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου του επιχειρηματικού είναι ακριβώς η έλλειψη λογοδοσίας παγκοσμίω. Τώρα, πέρα από την περιπλοκότητα των διαφόρων μορφών εργασία και των επιχειρηματικών μοντέλων, έχουμε πολλά νέα χαρακτηριστικά όπως αυτά που βλέπουμε και τα οποία αποτελούν παλαιές μεθόδους για την παράκαμψη των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων μέσω τεχνολογίας. Υπάρχουν ε, τρόποι όμως για να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε ας πούμε, να βασιστούμε στην εθνική νομοθεσία, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και στα διεθνή ε, πρότυπα όπως διεθνείς χάρτες, συμβάσεις κλπ. Επίσης είναι σημαντικό εδώ να ακολουθήσουμε και τη λογική. Το περασμένο μήνα η οργάνωσή μου είχε συμμετάσχει σε μια υπόθεση στον Μπαγκλαντές για την ασφάλεια στο χώρο εργασία ώστε να διασφαλίσουμε το ότι οι εργαζόμενοι ακριβώ, οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Ένα αυτοπασχολούμενο ε, στον τομέα των οικοδομών απεβίωσε μετά από ένα ατύχημα. Η επιχείρηση όμως δήλωσε πτώχευση. Δεύτερο παράδειγμα, εκμετάλλευση ανηλίκων. Ε, σε αυτή την περίπτωση είπε η επιχειρήση ότι κατά λάθο δήλωσε την ηλικία του στην ε, αίτηση αυτό ο εργαζόμενο. Μετά κάποια άλλα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν Μετά από συζητήσει που είχαμε στα μέλη των οργανώσεών μας. Για τους εργαζόμενου καταρχάς, οι ψευδοαπασχολούμενοι κατατάσσονται και αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με του ε, κανόνε ασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, ε, με τις επιθεωρήσεις εργασίας και του πόρου που διαθέτουν. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο και πιο πρακτικό ορισμό στην Ένωση για τον εργαζόμενο, ώστε να καλύψουμε όλου του εργαζόμενου, ιδιαίτερα αυτού που είναι ε, εργαζομένοι online στο ίντερνετ. Εμείς αυτό που προτείνουμε ως συνδικάτα είναι μια χωριστή κατηγορία που θα καλύπτει τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων που εργάζονται διαδικτυακά. Και νομίζω ότι αυτά που έγιναν πρόσφατα στο Μένο Βασίλειο πήγαν στη λάθο κατεύθυνση. Επόμενο σημείο, για του για τους εργοδότε, για του αυτοπασχολούμενου, θεωρούμε ότι υπάρχει μια σχέση εργασία και ότι το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι αντιστρέψιμο ώστε να πρέπει να, αποδείξει ο εργοδότης δεν πραγματικά απασχολεί τον εργαζόμενο. Μετά η διαμεσολάβηση για τις ε, διάφορες ε, πτυχές της λειτουργίας του, το ρόλο του εργοδότη. Θα πρέπει να το δούμε αυτό ώστε να το προσαρμόσουμε σε διάφορα φαινόμενα που υπάρχουν όπως οι υπηρεσία συνταγραφεία προσωρινής απασχόλησης και η περίπτωση υπεργολαβίας. Μετά, θα πρέπει να πούμε ότι όλο και πιο συχνά οι απασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι έχουν διάφορους, πέραν του ενός δηλαδή, εργοδότες. Εδώ θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται, να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να καταμερίσουμε την ευθύνη, ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων διασυνοριακά. Μετά χρειαζόμαστε επίση νομοθεσία για να επιβάλλουμε στους εργοδότες να συμβάλλουν στο κομμάτι που σας δικεί στην κοινωνική πρόνοια. Οπότε θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε το πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν όχι μόνο σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και στα συστήματα πρόνοιας στις περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος παρέχει διαφορετικό είδος υπηρεσιών. Μετά άλλο ένα σημείο βασικό για μας. Ανεξάρτητα από το καθεστώς εργασίας του αποσχολούμενου αυτοί θα πρέπει να καλύπτονται από πλήρη καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα ελάχιστη αμοιβή, ελάχιστου εκατότατου μισθού. Δεν είναι αποδεκτό να έχουμε, ας πούμε, ορομίστιο μία ώρα τη στιγμή που το ορομίστιο είναι 8 ευρώ την ώρα. Και επίσης πρόσβαση στην κατάρτιση και διαβιομάθηση. Μετά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Δικαίωμα εκπροσώπηση, δικαίωμα συμμετοχή σε συλλογικέ διαπραγματεύσει και εδώ ακριβώ θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι συλλογικέ διαπραγματεύσει αφορούν συνθήκε εργασία των εργαζομένων. Δεν έχουμε να κάνουμε με τι τιμέ των υπηρεσιών και των αγαθών, οπότε δεν είναι θέμα καθαρά ανταγωνισμού, γιατί αυτό πρέπει να καλύπτει και του αυτοαπασχολούμενου. Το δικαίωμα για συλλογικέ συμβάσει είναι ένα δικαίωμα καθολικό. Μετά χρειαζόμαστε μια ισχυρή επιθεώρηση εργασία με την ε, κατάλληλη στελέχωση. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ πώ οι επιθεωρήσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να συνεργαστούν διασυνοριακά ή θα μπορούσαμε ενδεχομένω να, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργία ενό πανευρωπαϊκού ε, ε γραφείου επιθεώρηση εργασία. Θα πρέπει να δούμε επίση και άλλα θέματα όπως η προσωρινή απασχόληση όπου υπάρχουν κενά και που, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινούν εργαζόμενους και να παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους για τις συλλογικές συμβάσεις και την ε, στην κοινωνική πρόνοια. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπουμε στις οικογένειες να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό είναι βασικό για την ίδια την ζωή των, και την ασφάλεια των εργαζομένων στο να υπάρχει κάποια σχετική προβλεψιμότητα και ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστέ οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπεί αμοιβή. Αυτό νομίζω αναπόσπαστο κομμάτι τη κοινωνία μα, Μετά για τι πλατφόρμες, πριν από 10 χρόνια η οργάνωσή μα είχε ζητήσει ο τομέα τη προσωρινή απασχόληση να Ελεχθεί. Σήμερα υπάρχουν ε, πλατφόρμες που θα πρέπει να συνεργαστούν με τα συνδικάτα ώστε να καλύψουμε αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να τα πράξουμε αυτά μαζί, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, αλλά και κοινωνικοί εταίροι νομίζω, όπως και εργοδότες, θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο Αυτά από μένα σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ε, καλά τα είπατε για συνδικαλιστής. Ε, γιατί ξέρω, σας το λέω. Γιατί ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε κατόπιν τον στην Βρέκε από τον ΩΣΑ. Σας ακούμε. Um, um, Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ. Θα μιλήσω για την κοινωνική προστασία κυρίως στην συνεργατική οικονομία. Πρώτον, η συνεργατική οικονομία παραμένει σχετικά μικρή. Δεν με δίστανται, κάποιοι λένε 0,5, άλλοι λένε 5%, αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί ως προς τους, ε, το, το, το, τι είναι συνεργατική οικονομία κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις ε, περιπτώσεις ε, οι εκτιμήσεις κρατήνουν σε κάτι πολύ μικρό. Παρ' όλα αυτά, η τάση είναι αυξητική, τη βλέπετε δεξιά. Βλέπετε τις ε, πέντε βασικές πλατφόρμες, όπως το Amazon, το p κλπ. Το Guru εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον αλλά και η προσφορά αυξάνονται ταχύτερα. Το σημαντικό προκειμένου είναι ότι προς το πάνω δεν ξέρουμε. Να δείσουμε λίγο στα τυφλά. Οι περισσότερες έρευνες στα νοικοκυριά, στου απασχολημένου κλπ. δεν μετρούν την συνεργατική οικονομία. Θα χρειαζόμαστε μια στοχευμένη έρευνα. Επίσης, τα φορολογικά στοιχεία δεν μας βοηθούν επαρκώ. Οι άγνωστοι λοιπόν είναι πολλοί εδώ. Ποιοι είναι καταρχήν αυτοί οι εργαζόμενοι, τι κάνουν, πού δουλεύουν, πού παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αποτελεί αποτέλεσμα επιλογής η απασχόληση αυτή. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, είναι κύρια εργασία τους, είναι δευτερεύουσα, πώς βγάζουν και ούτω καθεξής. Όλα αυτά για να τονίσω για μια φορά ότι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για την συνεργατική οικονομία και ότι χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν έχει τη ώρα να πάρουμε αποφάσεις πολιτικής. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα με την έννοια ότι το πρόβλημα δεν είναι απομονωμένο. Ε, τα ζητήματα αυτά υπάρχουν γύρω μας εδώ και δεκαετίες. Για να δούμε τους μέσους όρους του ΟΣΑ. Πάνω από 15% των ανθρώπων είναι αυτοπασχολουμένοι. 16% δουλεύουν σε βάση μερικής απασχόλησης και 13,5% σε προσωρινή απασχόληση. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν με μη συμμερικές μορφές εργασίας. Μη μισθωτή σχέση δηλαδή. Πολλά από τα προβλήματα που συζητούμε εδώ είναι προβλήματα τα οποία αφορούν και την συνεργατική οικονομία. Όπως είπα, θα μιλήσω για κοινωνική προστασία. Έχω φέρει μερικά γραφικά εδώ, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε, όμως προσέξτε το εξή. Στην κοινωνική προστασία γνωρίζουμε ότι πρέπει να διακρίνουμε την νομοθεσία που καλύπτει πολλούς εργαζομένους, αυτούς που έχουν πρόσβαση τουλάχιστον, αξιοποιούν την νομοθεσία. Πρώτη για νομοθεσία που είναι λιγότερο γενναιόδορη θα έλεγα προς τις νέες μορφές εργασίας. Ανεξάρτητους ε, αυτοπασχολούμενους ε, οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείονται. Σας δείχνω εδώ μερικές ε, χώρες και τις παροχέ που εξασφαλίζουν σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην συνεργατική οικονομία είναι αυτοπασχολουμένοι. Λοιπόν, το πράσινο, το χαμόγελο, σημαίνει πλήρη πρόσβαση στις παροχές του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το ανοιχτό πράσινο σας λέει πρόσβαση, αλλά εθελοντική, σε θελούσια βάση. Το πορτοκαλί μας λέει ότι στη συγκεκριμένη χώρα υπάρχει πρόσβαση, αλλά μερική και μόνο. Οι κανόνες δηλαδή διαφέρουν για τη συνεργατική οικονομία ή οι παροχές είναι χαμηλότερες και το κόκκινο σημαίνει καμία παροχή. Θέλω να πω τα εξή τώρα. Όσον αφορά την ε, σύνταξη, αναπηρία, επιδόματα πατρότητες, μητρότητες κλπ. Τα πράγματα δεν είναι άσχημα, αλλά διαφέρει πολύ η κατάσταση όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε τα θέματα ατυχημάτων και ενεργεία. Η Σουηδία, βλέπετε, είναι μια χώρα, δηλαδή, είναι χώρες που πηγαίνουν πολύ καλά σε όλου του τομεί, υπάρχει σχεδόν εξομοίωση, όμω σε άλλες χώρες υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αυτούς του εργαζομένου, λοιπόν, θα έπρεπε να του καλύψουμε. Αυτή είναι η νομική πτυχή του προβλήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πράξη όμως, ακόμη και αν θεωρητικά έχεις πρόσβαση σε αυτές τις διατάξεις, μπορείς να τις αξιοποιήσεις. Γιατί, Γιατί κάποιοι κανόνες δεν αποδίδουν στην πράξη. Ε, λόγω εισφορών, λόγω διάρκειας απασχόλησης κλπ. Στην πράξη λοιπόν κάποιοι δεν έχουν κοινωνική προστασία. Και δούμε μερικά παραδείγματα από μια τελευταία έκθεση της Κομισιόν. 55% των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, ε, δεν έχουν δικαίωμα σε επίδομα ανεργία. 38% δεν έχουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενεία και 46% των αυτοαποσχολημένων γυναικών, μισέ δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα σε επίδομα μητρότητα. Πολλέ φορέ γιατί δεν πληρούν κάποια κριτήρια ή επειδή πολλέ φορέ για λόγου φορολογικού δουλεύουν απλά μαύρα. Στην άτυπη οικονομία. Πώ θα τα διορθώσουμε λοιπόν όλα αυτά. Πρώτον, πρέπει να διορθώσουμε το σύστημά μας και μπορούμε να κάνουμε πολλά προκειμένου. Πρώτον, γνωρίζουμε στη συνεργατική οικονομία ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο προς το παρόν ότι υπάρχει ένα θέμα με την ταξινόμηση των υπαλλήλων, την κατηγορηποίησή τους είτε την κάνουν οι εργαζόμενοι είτε οι εργοδότες και εδώ υπάρχουν πολλά κίνητρα νομοθετικά αλλά και φορολογικά, να περάσει ο κίνδυνος στους ώμους του εργαζομένου. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει λοιπόν τις διαφορές αυτές να τις εξαλείψουμε, να εξαλείψουμε τα κίνητρα κακής καταχρηστικής των εργαζομένων. Επίσης υπάρχουν παραθυράκια και ασάφειες. Ο Λακρίγκερ στις ΗΠΑ το είπε. Η κατηγοριοποίηση αυτών των υπαλλήλων μοιάζει με τετραγωνισμό του κύκλου πολλές φορές. Ύστερα προκύπτουν νέες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα δεν λύνει ούτε τα νομοθετικά, ούτε τα προβλήματα ταξινόμησης κατηγοριοποίησης των εργαζομένων. Ακόμα και εκεί που οι κανόνες είναι σωστοί, πρέπει να εφαρμόζονται. Και αυτό λέω εδώ. Οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται, το ξαναλέω, και αυτό σημαίνει κυρώσεις όπου είναι απαραίτητο. Σε πολλές χώρες δεν προβλέπονται κυρώσεις καθόλου ή κάποιες αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται στην πράξη τελικά. Όσο αφορά του εργοδότε γιατί εδώ πρέπει να ρίξουμε το βάρο μα. Ε, Μπορεί να γίνουν πολλά, αλλά τα θέματα είναι και θέματα των εργαζομένων. Πολλές φορές η καποιε αποφασει δικαστηριων δεν εφαρμοζονται στην πραξη τελικα οσον αφορα του εργοδοτε γιατι εδω πρεπει να ριξουμε το βαρο μα μπορουν να γινουν πολλα αλλα τα θεματα ειναι και θεματα των εργαζομενων πολλε φορε η εργασια ειναι αδηλωτη για φορολογικού λόγου. Πολλέ πλατφόρμε πρέπει να μπουν μέσα στο φορολογικό σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απ' έξω. Τέλο, σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα. Ανεξαρτήτω κατάταξη εργαζομένων και ανεξαρτήτω των φορολογικών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζομένοι αυτοί έχουν επαρκή κοινωνική προστασία. Θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τι νομοθετικέ, κανονιστικέ πτυχέ, αλλά και τα πράγματα στην πράξη. Πώ μπορούμε να επεκτείνουμε την κοινωνική ασφάλιση και σε αυτέ τι ευέλικτε μορφέ εργασία, αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε. Σε μερικέ περιπτώσει Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικού μηχανισμού για του αυτοπασχολουμένου είτε στην τέχνη, στην γεωργία κλπ. ώστε τελικώ οι άνθρωποι αυτοί να έχουν προστασία. Και τέλο, μπορούμε να συμπληρώσουμε τα υφιστάμενα σχήματα, έστω και χωρί ε, εισφορέ εργαζομένων, για να υπάρχει δίκτυο προστασία. Όσον αφορά την ουσιαστική πρόσβαση, εάν κάποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσον αφορά τι κοινωνικέ παροχέ υπάρχει τέλο πάντων ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε είτε με υφιστάμενους μηχανισμού είτε με νέου. Αρκεί φυσικά να πληρούνται κάποια κριτήρια από την πλευρά των εργαζομένων. Και τέλο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι φορητά. Πρέπει να έχει φορητότητα όταν αυτοί περνούν από τη μία μορφή εργασία στην άλλη, να μην χάνουν την προστασία. Θα αφιερώσω τα τελευταία λεπτά που έχω στη θέση μου για να συζητήσω το θέμα της αντικατάσταση, ή της υποκατάστασης, αν θέλετε, των εφισταμένων μηχανισμών κοινωνικής προστασίας με νέους. Σε κάποιες χώρες οι κυβερνήσεις πειραματίζονται. Το συζητούσαμε και στον ΩΣΑ πρόσφατα και προσπαθούμε να δούμε πόσο εφικτό θα ήταν ένα ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα. Υπάρχουν πολλά θετικά εδώ. Πρώτον είναι απλό, γιατί όλοι προστατεύονται. Είναι λιγότερο πατερναλιστικό, λίγο κυδεμονευτικό, γιατί ε, όλοι παίρνουν το ίδιο. Και τρίτον, ε, εξελίφθεται το στίγμα κάποιου που είναι σε ένδια και χρειάζεται κοινωνική προστασία. Υπάρχουν φυσικά και πολλά εμπόδια στην εφαρμογή του. Το πρώτο και το προφανές είναι το κόστος. Αν αντικαθιστούσε κανείς τα επιδόματα. Το, το, το στέγης και αναπηρία με ένα βασικό εισόδημα, βασικό εγγυημένο εισόδημα, το κόστος δεν θα ήταν υψηλότερο και όλοι θα ήταν καλυμμένοι. Και όλοι βεβαίω θα ήταν πάνω από το κατόφλι τη φτώχεια. Γι' αυτό φυσικά θα χρειάζονταν περισσότερα χρήματα και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι και κάποιε άλλε πηγέ. Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρέπει να πω ότι σίγουρα κάποιοι θα χάσουν και κάποιοι θα κερδίσουν εάν εφαρμοστεί. Θα κερδίσει σε τάξη, θα χάσουν ίσως αυτοί που αυτή τη στιγμή πράττουν πολλαπλά επιδόματα, για παράδειγμα μονογονικές οικογένειες. Θα σταματήσω εδώ, απλώς να σχολιάσω το εξή ε, αφιέρωσα την ομιλία μου στην κοινωνική προστασία, αλλά ε, υπάρχουν και θέματα ε, δεξιοτήτων ε, και το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη συζήτηση για την κατάστασή τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Με το ελάχιστο εισόδημα έρχεστε βεβαίως στην έκθεση που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Νομίζω να μπορούσατε να συνεισφέρετε και εκεί. Οπότε παρακαλώ τον καθηγητή Μαρτίν Ρίσακ από το Ινστιτούτο Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που υπάρχουν τόσο πολλοί διερμηνείς και θα μιλήσω γερμανικά. Ε, λοιπόν, τίτλο έχω βάλει εδώ πέρα η οικονομία των πλατφορμών, αλλά όπως είπε και η συνάλφος, η ορολογία αυτή αποκλίνει από την επίσημη ορολογία της Ένωσης που μιλάει για συνεργατική οικονομία και ακριβώς ε, όταν δεν έχει επικρατήσει μία ενιαία ορολογία ε, υπάρχει ένα ζήτημα και βεβαίω όταν μιλάμε για μια συνεργατική οικονομία ακούγεται πάρα πολύ θετικό όταν μιλάμε για οικονομίες πλατφόρμας ε, είναι κάτι το ουδέτερο, όχι αρνητικό. και ε, υπάρχει ακριβώς η έννοια του ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι. Όταν μιλάμε για γι, η οικονομία του gigabyte επίσης σημαίνει κάτι άλλο. Και ότι υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις. Λοιπόν, να δούμε το φαινόμενο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξή. Ε, κατά κανόνα όταν μιλάμε για νέους τρόπους εργασίας, για καινοτομία για όλα αυτά. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι πράγματι νέα και καινοτόμα και πολύ θετικά. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που είναι κοινό και αφορά τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης. Έχουμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που λέγεται επισφάλεια. Βεβαίω δεν είναι και αυτό κάτι το καινούριο. αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα αρνητικά κυρίως επικεντρώνονται στους εργαζόμενους. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές μορφές ε, απασχόλησης που ε, μας απασχολούν κυρίως. Υπάρχουν δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι οι οποίοι ενσωματώνονται σε έναν μεγαλύτερο ε, οργανισμό με μια πιο ευέλικτη σχέση εργασίας είτε μιλάμε για μερική απασχόληση, είτε για χρονικά περιορισμένη σύμβαση, είτε με άλλες μορφές ε, τέτοιες. Και βεβαίως η οικονομία αυτή είναι μια συνέχεια αυτής της μετατόπισης ε, του ρίσκου τελικά στους εργαζόμενους. Και το ρίσκο αυτό έχει τη μορφή της μη απασχόλησης. Και βλέπουμε ακριβώς ε, ότι αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στα συμβόλαια τα ορομίσθια, όπου έχει ο άλλος την υποχρέωση να είναι μονίμως ε, διαθέσιμος και θα, ε, θα έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει αυτή η οικονομία μόνο όταν ισχύουν δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι όταν θα υπάρχει ένα σε αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων που πράγματι ζητάνε την υπηρεσία και βλέπουμε ότι ένα από τα καινοτόμα στοιχεία είναι ότι χρησιμοποιούν και δημιουργούν ένα μεγάλο τέτοιο πλήθος ε, δυνητικών ε, πέλατων. Γι' αυτό ακριβώς απαιτείται όσο δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία από τους εργαζόμενους. Το δεύτερο που δεν αναφέρθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την ψηφιακή φήμη. Δηλαδή ότι υπάρχει ο έλεγχος ποιότητας, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ε, για αυτούς οι οποίοι όντως θα ζητήσουν αυτήν την ε, υπηρεσία. Και αυτό τελικά αντικαθιστά την σχέση της απασχόλησης. Και ε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την ψηφιακή φήμη και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν μιλάμε για άτομα τα οποία υποτίθεται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Λοιπόν, να αναφέρω τώρα δύο πράγματα. Το ένα είναι από ένα άρθρο. Προ ίντερνετ ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάποιον, να καθίσουμε μαζί του 10 λεπτά να δουλέψει για μας και μετά να τον απολύσουμε μετά από 10 λεπτά. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει με την τεχνολογία. Αυτό νομίζω μας δείχνει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τώρα το άλλο. Αν δούμε το εργατικό δίκαιο αφενός και την κοινωνική ασφάλιση και από την άλλη την εργατική οικονομία έχουμε διάφορα προβλήματα. Το βασικότερο, το βασικότερο πρόβλημα είναι το θέμα της κατάταξης. Τα άτομα αυτά είναι όντως αυτοαπασχολούμενοι όπως ισχυρίζονται οι περισσότερες πλατφόρμες ή έχουμε σχέσεις εξαρτημένης εργασίας. Ε, πρέπει να διακρίνουμε, δηλαδή όταν μιλάμε για το Uber έχουμε μια ομάδα τέτοια. Υπήρχε και μια απόφαση νομίζω του σχετικού δικαστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλλο είναι όταν έχουμε κάποια εικονική εργασία που μοιράζεται σε πάρα πολλούς ε, όπως ε, με τις διάφορες πλατφόρμες της Amazon ή μέσω του Clickworker, του Upwork κτλ. Εκεί πέρα πράγματι είναι ένα ερώτημα και που μπορεί βεβαίως κανείς να προσφύγει όταν εργάζεται σε έναν εικονικό χώρο. Και βεβαίως ε, το άλλο αφορά το θέμα παραδείγματος χάρη ατόμων τα οποία βοηθούν στο νοικοκυριό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιος είναι τελικά ο εργοδότης όταν έχουμε, παραδείγματο χάρη, τριμερείς ε, συμβάσεις. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες παρόμοιες σχέσεις εργασίας από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε. Από την άλλη υπάρχει στην θεωρία η λεγόμενη λειτουργική έννοια του εργοδότη, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος πράγματι επιτελεί τον ρόλο του εργοδότη, ποιος έχει τις ευθύνε, ποιος είναι υπεύθυνος παραδείγματο χάρη για να τηρήσει τα του βασικού μισθού της κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Λοιπόν, ποιες στρατηγικές υπάρχουν. Θεωρώ πως ε, ε, υπάρχουν τρεις ε, κύριες στρατηγικές. Η πρώτη αναφέρθηκε, το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μία ενδιάμεση κατηγορία, δηλαδή εάν ε, μπορούμε να τους κατατάξουμε στις υφιστάμενες κατηγορίες που είχαμε. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό. Περισσότερες χώρες ε, αναφέρουν Παραδείγματο χάρη ε, το ότι ήδη στην Γερμανία στο Μεσοπόλεμο υπήρχε μια τέτοια ενδιάμεση κατηγορία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά νέα αυτή η κατηγορία, αλλά παρόλα αυτά είχε εμφανιστεί πριν από την συνεργατική οικονομία. Να σας υπενθυμίσω ότι υπήρχε εδώ πέρα και μια λευκή βίβλωση για τον εξυγχρονισμό του εργατικού δικαίου και εκεί πέρα είχε προταθεί μια ενδιάμεση ε, κατηγορία την οποία θα μπορούσαν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο, επίσης, ε, το οποίο ε, αναφέρει και ο από το Συνδικάτο, είναι ότι θα πρέπει να επανακαθορίσουμε την έννοια του εργαζόμενου, το οποίο βεβαίως είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται προστασία από τους δύο συμβαλόμενους Εκεί πέρα υπάρχει λεγόμενη ε, φόρμουλα Lowry Bloom ε, για να το καθορίσουμε αυτό. Αλλά το θέμα βεβαίως ε, μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο πολύ θέμα προστασία, αλλά περισσότερο ελευθερία, ειδικά όταν μιλούσαμε για τον δημόσιο τομέα. Αλλά δεν νομίζω πλέον να υπαρκούν αυτά τα πράγματα για τις ε, τωρινές ε, εργασιακές σχέσεις. Η τρίτη δυνατότητα είναι να πούμε ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή ρύθμιση, μια οδηγία παραδείγματο χάρη για το crowdwork. Αναφέρθηκαν ήδη κάποιες δυνατότητες. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε είναι να υπάρχει το βάρος της απόδειξης το οποίο θα πέφτει στην πλατφόρμα. Να πρέπει η πλατφόρμα δηλαδή να αποδείξει ότι κάποιος δεν είναι υπάλληλο, δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας. Θεωρώ πως η διαφάνεια, η πληροφόρηση έχει εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση πληροφόρηση και να υπάρχουν κάποιοι όροι των συμβάσεων που θα απαγορεύονται. τέλο, πάρα πολύ σημαντικό, αφορά τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις ε, και συμβάσεις. Έχουμε και το άρθρο 101 της συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά ειδικά τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε πράγματα τα οποία ισχύουν ήδη όταν μιλάμε παραδείγματο χάρη για την απόφαση του δικαστηρίου Κούνστεν που αφορά τους ψεύδο αυτοαπασχολούμενους, τα λεγόμενα μπλοκάκια παραδείγματο χάρη. Τώρα, το θέμα είναι ποια είναι η δυνατότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ποιος ε, περιλαμβάνεται, στο πεδίο προστασίας. Το δεύτερο είναι πώς θα οργανώσουμε την κοινωνική ασφάλιση όταν υπάρχουν παραδείγματο χάρη αυτές οι κατακρεματισμένες εργασιακές σχέσεις και το τελευταίο βέβαια που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν θα πάμε, εφόσον πηγαίνουμε προς αυτές τις ε, μορφές ε, εργασίας ε, να δούμε τι σημαίνει αυτό τελικά για τα συστήματα κοινωνική ε, ασφάλισης ε, και πώς ε, θα δημιουργείται το εισόδημα και το κεφάλαιο το οποίο απαιτείται για την κοινωνική ασφάλιση. Σας ευχαριστούμε και σας κύριε καθηγητά. Περνάμε λοιπόν στον πρώτο κύριο της συζήτησης. Να δούμε πρώτα απ' όλα τους συντονιστές. Πρώτος ο Χάιντς Μπέκερ για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω στο βήμα αγαπητέ φίλε. Ήταν ευχαριστή εκπλήξη. Να ευχαριστήσω τώρα τους τέσσερις ε, ομιλητές μας. Έχουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου όλα όσα λέμε και περιγράφουμε κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικό κράτος ε, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της συνεργατικής οικονομίας και παρόλο παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι ακόμα σαφής η όρη, είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη δράσης. Ε, και δεν θέλω να κρύψω πως ε, η κατάταξη όλων αυτών των μορφών εργασίας ε, και απασχόλησης θα πρέπει να γίνει εντός της κοινωνικής οικονομίας αγοράς και όπου δεν υπάρχει σαφήνεια θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες νέες ρυθμιστικές προτάσεις. Γιατί ρυθμιστικές προτάσεις, γιατί δεν έχουμε στους περισσότερους από αυτούς τους τομείς νομοθετική αρμοδιότητα. Δεν μπορούμε να ε, παρέμβουμε άμεσα, αλλά ότι πρέπει να διδαχθεί η επιχειρηματικότητα, ότι πρέπει να υπάρχει το ωράριο, ο χρόνος ε, εργασίας, ανεξαρτήτως της ε, μορφής της εργασίας. Θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι κάτι στο οποίο μπορεί να παρέμβει και είναι η κατάλληλη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε εμείς δηλαδή να αναπτύξουμε τις ε, καταλληλότερες έννοιες για να καλύψουν αυτές τις νέες μορφές ε, απασχόλησης για να μην έχουμε ακριβώς ε, φαινόμενα τα οποία είναι απαράδεκτα. Και να ότι δεν έχουμε πράγματι νομοθετικές αρμοδιότητες, αλλά να μην υποτιμούμε τον soft την ήπια e ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά αν εγκρίνουμε κάτι με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ, Χάιντς, και για την προσωπική σας παρατήρηση. Τώρα, Γιώργη Σούστερ, ο οποίος ήταν ο εισηγητής για την ε, θέση που ανέφερα Τη επιτροπή μας που εντωμεταξύ εγκρίθηκε και από την Ολομέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις ε, ομιλίες αυτές με τις οποίες συμφωνώ σε μεγάλο μέρος. Να πω όμω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ε, λέτε ότι δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε αυτά γιατί είναι καινούργια. Εγώ δεν βλέπω τι είναι το τόσο καινούριο. Και η παραδοσιακή οικονομία έχει πάρα πολύ διαφορετικές μορφές εργασίας. Ε, αν δούμε πώς είναι, πόσα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και επιλέξαμε ακριβώς εμείς τον όρο οικονομία των πλατφορμών γιατί όλοι οι άλλοι όροι αποκρύπτουν το φαινόμενο. Για να δούμε λοιπόν. Είναι πραγματικά καινούρια όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι το καινούριο υπάρχει στο Uber. Ε, υπήρχαν πάντα ε, η δυνατότητα στη Γερμανία να νοικιάσεις μία λιμουζίνα με σοφέρ. Εντάξει, η διαφορά είναι ότι δεν παίρνεις τηλέφωνο, αλλά μπαίνει στο ίντερνετ. Αλλιώ δεν υπάρχει κάτι το καινούριο. Οπότε δεν ξέρω γιατί αποκλίνουμε από την κανονική ρύθμιση των επιχειρήσεων ταξί ή των αυτοκινήτων με σοφέρ. Επειδή η μόνη διαφορά είναι ότι δεν παίρνεις τηλέφωνο ας πούμε και γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, βασικό θέμα να για να ρυθμίσουμε είναι το ερώτημα ε, μήπως υπάρχει αναλογία με τα κλασικά επιχειρηματικά μοντέλα επειδή διαφέρει λίγο η τεχνολογία. Πράγματι έχουμε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό ναι, της αγοράς αλλά δεν ξέρω αν το ουσιαστικό είναι αν διαφέρουν κάποια χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι βασικές αρχές. Ε, έχουμε κάποια ζητήματα που υπάρχουν στην παραδοσιακή οικονομία. Οπότε κύριε Μπέκε είπατε πως είναι όλοι αυτοί σχεδόν όλοι αυτοαπασχολούμενοι. Και από πού βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, γιατί έτσι λέει η πλατφόρμα και άρα δεν χρειάζεται να τους ε, ασφαλίσει. Όχι. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Και δεν βλέπω πραγματικά, ε, όπως σας είπα, τι είναι το πραγματικά καινούριο και πώς αιτιολογούμε ότι η άνθρωποι είναι όντως αυτό που ασχολούμαι. Σας ευχαριστώ. Α, είναι δύο λεπτά παρακαλώ συντονιστές, ξέχασα να το πω. Άνθια Μακιντάιρ δεν είναι εδώ. Οπότε έχουμε τώρα τον Ενίκη Καλβεζαμόνου, ούτε αυτός είναι εδώ. Από την ΚΟΕ. Α, η Τάνια Γκονζάλης. Ε, βέβαια, το χαρτάκι τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπό τον όρο οικονομία διαμοιρασμού, που είναι ένας ωραίος ελκυστικός όρος, φαίνεται ότι φτάνουμε σε εργατικές ε, σχέσεις όπου δεν υπάρχει καν εργασία, ούτε καν προσπαθεί κανείς να δουλέψει. Υπό αυτόν τον όρο λοιπόν νομίζω ότι φαίνεται να κρύβονται σημαντικές μεταβολές όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις και τις παραγωγικές σχέσεις. Και όλο και περισσότερο περιλαμβάνει αυτός ο όρος ε, ποικίλε υπηρεσίες, μεταφορών, καθαριότητας και πολλές άλλες υπηρεσίες που φαίνεται ότι όλο και περισσότερες υπηρεσίες θα ενταχθούν στην ομπρέλα αυτή της ε, συνεργατικής οικονομίας διαμοιρασμού, όπου οι εργαζόμενοι δεν είναι πια εργαζόμενοι, αλλά είναι συνεργάτες. Δηλαδή, δεν κάνουν πια μια δραστηριότητα με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή, αλλά κάνω αυτή την δραστηριότητα επειδή ακριβώς και εδώ την κάνω εθελοντικά και με τρόπο έτσι συνεργατικό. Να δούμε όμως πώς έχει η πραγματικότητα. Θα δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, οι εργαζόμενοι του Deliveroo που απεργούν, οι αναβάτες του Deliveroo πρέπει να πληρώσουν την ασφάλισή τους, το ποδήλατό τους, το τηλεφωνό τους. Αν πέσουν και έχουν κάποιο τραυματισμό, δεν καλύπτονται από την επιχείρηση. Γιατί θεωρείται εκτός εργασίας το ατύχημα. Ελέγχονται μέσω GPS στην ουσία εργάζονται με μπλοκάκι, με βάρδιες τριώρες, 4-20 ευρώ αναπαραγγελία και δεν αμείβονται ανά ώρα, αλλά αναπαραγγελία. Συνήθως δύο παραγγελίες την ώρα. Διαμαρτύρονται λοιπόν ότι για το ότι η επιχείρηση θεωρεί ότι αυτή η εργαζόμενοι είναι στην ουσία αποσυνδεδεμένοι. Και τι είναι, ποιο είναι το νέο εδώ πέρα το κοινοτόμο. Το νέο είναι εδώ ότι μπορούμε στην ουσία να παρακάψουμε οποιοδήποτε εργασιακό νόμο ή νόμο κοινωνικη περιθαλψής ή πρόνοιας με αυτές τις νέες μορφές εργασίας. Υπ' αυτή λοιπόν την άποψη υπήρχε μια πρόταση για να γίνει μια διαφοροποίηση σε σχέση με την ορολογία. Δεν είναι το ίδιο η συνεργατική οικονομία με την οικονομία των πλατφορμών. Και κατά λίγο υπήρξε και η πρόταση για δυνατότητα κοινωνικών εισφορών ώστε να προσαρμόσουμε την αγορά εργασίας και τους κανόνες και να αντιμετωπίσουμε αυτή την άτυπη μορφή εργασίας, την ανασφαλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Εξαιρετικές εισηγήσει με πολλές χρήσιμες σκέψεις. Θα ήθελα να εμβαθύνουμε στο εξή, στην διασυνοριακή διάσταση. Γιατί αυτό κάτι, κάτι πρέπει να μας πει εδώ. Και νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στις δικές μας αρμοδιότητες διότι συζητούμε θέματα συντονισμού, διασυνοριακού συντονισμού συστημάτων κοινωνική ασφάλισης. Λοιπόν, ανεξαρτήτω τώρα των ορισμών, περί τι είναι αυτοπασχολούμενος, από τη μία χώρα στην άλλη, είναι δεδομένο, θεωρώ, ότι υπάρχουν κενά. Για να το συζητήσουμε αυτό θα ήθελα, παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα τη αυτοπασχόληση, άκουσαμε διάφορα από την Κομισιόν, έχουμε συζητήσει και εμεί το θέμα εδώ κατά επανάληψη, Ακούμε για την επιχειρηματικότητα, λέμε ότι πρέπει να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα. Αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο να προτείνεται αλφαγιώτα, ως λύση στο πρόβλημα της ενεργείας. Και ρωτώ, τα κράτη-μέλη κάνουν κάτι προκειμένου στο φορολογικό, στην κοινωνική ασφάλιση. Έχουν κατανοήσει τα προβλήματα πραγματικά προσπαθούν να τονώσουν αυτή τη μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να περάσουμε στο σύστημα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν συστήματα που τελικώς παρέχουν προστασία στους εργαζομένους ή πάμε όλοι για το γκρεμό. Θα βρεθούμε όλοι χωρίς σύνταξη κάποια στιγμή. Ακούστηκε ότι κάποια κρατημέλη προσφέρουν αρκετά ικανή προστασία. Για να δούμε τι έχουν πετύχει αυτά τα κρατημέλη. Πώς το κατάφεραν. Πώς το εφαρμόζουν στην πράξη και να το συγκρίνουμε με την κατάσταση σε άλλες χώρες μέλη. Αυτό νομίζω θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Γιατί κατά τα άλλα μιλήσαμε για τη σχέση ισχύω στον ρόλο του πελάτη που με την ευκαιρία είναι άλλο ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε ξεχωριστά πώς εκπαιδεύουμε τους ε, πολίτες, τους καταναλωτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας ξανακούμε εδώ. Σας βλέπω σε φόρμα μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο και ευχαριστώ τους προλαλήσαντες. Συζητούμε ένα νέο θέμα. Και χαίρομαι που συζητούμε μια μεγάλη μετάβαση, μια σημαντική εξέλιξη από την συμβατική στην συνεργατική οικονομία. Με σκοπό κερδοσκοπικό. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή είναι ταχύτατη, αυτή τη νέα οικονομική δραστηριότητα, Απουσιάζει η νομοθεσία εδώ, απουσιάζουν οι κανόνες. Και εδώ να συζητήσουμε παρακαλώ το εξή. Θεωρούμε ότι οι κανόνες όσοι υπάρχουν δεν εφαρμόζονται. Η κοινωνία μας με την αυτοματοποίηση μεταμορφώνεται και μελέτες δείχνουν ότι σε πρώτη φάση θα χάσουμε θέσεις εργασίας. Πολλές θέσεις εργασίας. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό θα αφορά μόνο το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Τα μπλε κολλάρα, όπως λέγαμε παλιά στην ε, Γαλλία. Εδώ βλέπω παράκαμψη των κανόνων μεταξύ αυτών και της κοινωνικής προστασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι μορφές αυτές εργασίας εκφεύγουν, διαφεύγουν από την υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Είναι η μεταμόρφωση της κοινωνικής προστασίας. Οι νέες θέσεις εργασίας σίγουρα προσφέρουν ελευθερία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι Όμω ακόμα και η μισθωτή αυτών των αλυσίδων είναι ένα μικρό συμπλήρωμα το οποίο δεν αμείβεται καν καλά. Και αισθάνεται μάλιστα, ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο σημαντικό, ε, ότι οι θέσει εργασία αυτέ είναι ιδιαίτερε προσωρινέ όπω την Uber. Τι γίνεται όμω με του καταναλωτέ. Το μοντέλο είναι καινούριο. Εκεί ανταγωνιστικά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Για να δούμε η Ευρώπη θα μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη, τα οποία πολλές φορές σε διμερές επίπεδο με διάφορες διεθνείς συμφωνίες καταφέρνουν να ξεφεύγουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην συζήτηση. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 10 και 25. Προσπαθούμε λοιπόν να τα δούμε όλα. Αν τηρήσουμε το χρόνο θα τα καταφέρουμε. Άνες Σάντερ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους τέσσερις προσκεκλημένους εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με αυτή τη νέα μορφή οικονομίας και αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης. Για κάποιες ε, περιοχές αποτελούν ένα πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για κάποιες κατηγορίες όπως ανθρώπων όπως οι φοιτητέ που χαίρονται που έχουν ευκαιρίες εργασίας ή κάποιε και βοηθούς κλπ συγγνώμη, οικοκυρές κλπ. Αλλά όπως υπόθηκε, υπάρχουν και προβλήματα σε σχέση με αυτές τις μορφές εργασίας. Υπάρχουν καταχρήσεις που θα πρέπει βεβαίως να αντιμετωπίσουμε επειδή επιφέρουν κινδύνους ε, στην υγεία και την ασφάλεια. Νομίζω ότι οι τέσσερις εισηγητές αλλά και οι συνάδελφοι υπογράμμισαν ότι σήμερα παραμένουν πολλά ερωτήματα από ότι απαντήσεις που έχουν δοθεί. Εγώ θα ήθελα να μάθω πώς θα μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία, ώστε καλύτερα να κατευθύνουμε τις πολιτικές. Και άλλο ένα ερώτημα. Το είπατε κι εσείς, κύριε Ρισάκ, εξάλλου. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε καταρχάς. γιατί στις περισσότερες χώρες μη υπάρχει σήμερα καθεστώς απασχολούμενο ή αυτοαπασχολούμενο. Μήπως όμως πρέπει να κάνουμε νέους νόμους, να κάνουμε οδηγίες ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απλά και μόνο για να ενισχύσουμε ή ενδεχομένως για να ενισχύσουμε μόνο τις ε, εθνικές νομοθεσίες που αφορούν αυτά τα καθεστώτα εργασίας, ιδιαίτερα των αυτοαπασχολουμένων που ποικίλουν από χώρα σε χώρα της Ένωσης. Οπότε αυτά είναι τα ερωτήματα. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε πού, σε ποιες περιπτώσεις και πότε. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας παχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Νομίζω πολλά θέματα είναι ακόμα ανοιχτά. Και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσουν. Όπως είπε ο η το θέμα είναι επίσης ε, το σύστημα της συλλογής δεδομένων. Ε, κινούμαστε σε ένα πεδίο που μπορούμε να διαμορφώσουμε μόνο αν έχουμε ε, δεδομένα. Το θέμα είναι ποιες δυνατότητες έχουμε να τα διαμορφώσουμε. και ενδιαφέρον ήταν αυτό το οποίο είπε ο κύριος από που βλέπουμε τις πράσινες ε, φατσούλες ε, αφορούσε κυρίως βορειοευρωπαϊκές ε, χώρες αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις νότιες χώρες είναι σύμπτωση τι είναι εν τω μεταξύ υπάρχει όπως και, όντως και το ζήτημα των ψεύτων αυτό Έχουμε κάποιες ε, εμπειρίες και κάποια στοιχεία ε, για το τι γίνεται ε, και σε αυτούς τους κλάδους και σε άλλους. Εδώ έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε ακριβώς συλλάβει και δεν ξέρουμε την έκταση του φαινομένου που σχετίζεται επίσης και με την παράνομη εργασία. Πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να αποφύγουμε και να ελέγξουμε την παράνομη εργασία. Νομίζω ότι Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να, να γίνει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Χέντρικλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τις παρουσιάσεις τους σήμερα το πρωί που διαφώτισαν τη συζήτηση και μας εμπλούτησαν. Από ό,τι βλέπουμε, οι χώρες μέλη οπωσδήποτε θα πρέπει να προστατεύσουν τους απασχολούμενους, τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνειδητοποιούν πια ότι έχουν δικαιώματα. Επειδή σε κάθε χώρα θα πρέπει για να αποφευθεί ακριβώς η εκμετάλλευση, θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας. Επίσης έχουν ρόλο εδώ και ισχυρό μάλιστα οι καταναλωτές Μιλούσαμε προηγουμένως για συνεργατική οικονομία, η οικονομία πλατφόρμας, που είναι αξιόλογες μορφές, αλλά και οι καταναλωτές και πάλι θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο εδώ και θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το ενδεχόμενο εκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σωστό να έχουν βεβαίως κοινωνικά δικαιώματα, να καλύπτονται, να έχουν κοινωνική πρόνοια και προστασία, να έχουν κατάλληλους μισθούς, αξιοπρεπείς μισθούς οι εργαζόμενοι. Και αν μια υπηρεσία είναι ευθυνή, ας πούμε οι υπηρεσίες ε, ταξί σε σχέση με τα παρουσιακά ταξί. Για τις παραδοσιακές μορφές αυτών των υπηρεσιών υπάρχει ένα παραπάνω κόστος, αλλά αυτό αφορά τη στήριξη των εργαζομένων και την κατάλληλη προστασία τους. Οπότε οι καταναλωτέ θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ακριβώς να ξέρουν ποια είναι η αξία των φθηνών υπηρεσιών. Υπάρχει ένα θέμα εδώ εκπαίδευσης. Επίσης η αυτοαπασχόληση, αν είστε αυτοαπασχολούμενος, έχετε την ελευθερία να παράσχετε αυτή την υπηρεσία σε όποιο θέλετε, αντί να δεσμεύεστε ε, με μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή εργοδότη. Οπότε χρειαζόμαστε και σε αυτό το τομέα νομίζω ένα κατάλληλο ορισμό. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο τον λόγο. Υπάρχει κάποιο. παρακαλώ. Μία σύντομη συμπλήρωση. Ξέχασα να τονίσω ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εδώ και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Ευχαριστώ. σε. Ευχαριστώ. Κάποιος να παραγγείλει πριν κλείσουμε κάτι. Λοιπόν, η ειδικοί τότε, για πέντε λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ, απαντήστε. Άντε και έξι λεπτά. Η κυρία Ντουέ πρώτη. Microphone, please. Oh, sorry. Pardon me again. Uh, yes, I think on... Ναι, σας ευχαριστώ για τα σχολεία σας και τους εμπειρογνώμας για τις εισηγήσεις. Ε, επανειλημμένα ακούμε την έκκληση για σαφήνεια και ακόμα να γίνεται λόγος για συζητήσεις που πρέπει να προχωρήσουν. Το άλλο σχόλιο για τη συνεργατική οικονομία ή την οικονομία πλατφόρμας και συμφωνώ ότι ο όρος συνεργατική μπορεί να προδιαθέτει στο ότι δεν γίνεται κάποια δουλειά, αλλά ο όρος είναι σημαντικός για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε συζητήσεις. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όταν θα αναζητήσουμε λύσεις όπως είπαν εδώ και οι υπηρεγνώμονές μας, για να βρούμε λύση σε μια ταχεία εξελισσόμενη μορφή οικονομίας. Ακούσαμε επίση και μια σοβαρή ισχυρή έκκληση για δεδομένα, περισσότερα στοιχεία. Πριν να αναπτύξουμε λοιπόν και να ζητήσουμε λύσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε τι γίνεται βασισμένη σε επιστημονικές μελέτες και στοιχεία που αφορούν στους εργαζόμενους. Όσον αφορά εμά την οργανώσή μας για τη συνεργατική οικονομία στην Ιρλανδία, εμείς θέλουμε να εισακούσουμε όλους τους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα της οικονομίας που πολύ συχνά λείπουν από συζητήσεις που, γίνεται, που γίνονται για αυτό το τομέα, παρόλο που είναι στην ε, πρώτη γραμμή αυτού του κλάδου. Επίσης ακούσαμε εκκλήσεις για σαφήνεια, ξαναλέω και συνοψίζω, σαφήνεια, περισσότερα επιστημονικά στοιχεία και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα από όλες τις χώρες μέλη για σαφήνεια όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κάλυψή τους. Δεν είναι απαραίτητα σημείο αποφυγής γιατί αυτοί οι εργαζομένοι καμιά φορά απλά και μόνο δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Αυτό δεν γίνεται συστηματικά, αλλά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ενημέρωση και πρόσβαση στην ενημέρωση. Εγώ λοιπόν σε αυτά θα περιοριστώ. Στη μεγάλη έκκληση για σαφήνεια, και για την ύπαρξη επιστημονικών δεδομένων, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις οικονομίες πλατφόρμας. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω, να έχουμε πρωτοβουλίες που θα ενημερώνουν τον κόσμο για τα δικαιώματά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα. Να ασχολήσω αυτό που είπε ο κύριος Μπέκερ. Να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία. Η τεχνολογία έχει αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σήμερα τελευταία 200 χρόνια, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι εφαρμογή τη νομοθεσία. Γιατί για πολλά χρόνια οι επιχειρήσει έβρισκαν ε, ε, ωραίου τρόπου να φοροδιαφεύγουν, χρησιμοποιώντα βεβαίω άλλε μεγάλε επιχειρήσει που τι βοηθούσαν. αποσύροντας ευθύνες από τις επιχειρήσεις αυτές. Ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με αυτό άμεσα είναι η διασυνοριακή διάσταση που έθεσε η Τζιν Λάμπερτ και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ήδη το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας, στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε οι συνάδελφοι στον τομέα των οικοδομών σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυτά τα παραδείγματα όπου οι επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους από την Ρουμανία ας πούμε όπου είναι καλυμμένοι έχουν προνοια στην Κύπρο και δουλεύουν στην Ολλανδία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί όταν μιλάμε με τα μέλη των οργανώσεων μας, μας λένε ότι στην ουσία η νέα αγορά δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει. Δηλαδή η Ευρώπη δεν μας βοηθάει. Οπότε ας το δούμε συλλογικά αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε τι έγινε με το Brexit. Τα συνδικάτα δεν μπόρεσαν να πείσουν τα μέλη των συνδικάτων για το Brexit. Και αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε μόνο στον Βασίλειο αλλά και σε άλλες χώρες. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες και εδώ ακριβώς παραπέμπω στον Juncker όταν συζητάμε για τον κοινωνικό πυλώνα τα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει να έχουμε τέτοιες πολιτικές ώστε η νέα αγορά να βοηθά τους πολίτες. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο θέλετε, αλλά αυτό είναι το κυριότερο νομίζω. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τους αυτοαπασχολούμενους. Και πάλι πρόκειται για θέμα επιβολής της νομοθεσίας, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι εργαζόμενος με τον παραδοσιακό όρο και ποιος δεν είναι. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση λοιπόν να διακρίνουμε ποιος είναι εργαζόμενος και ποιο όχι. Δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε σε νομοτεχνικά ζητήματα, απλά και μόνο να κάνουμε μια πλήρη άκρηση τι είναι εργαζόμενος και τι δεν είναι. Επιχειρηματικότητα. Άλλο ένα θέμα που μου είναι προσφυλέ. Αν ω εργαζόμενος δεν μπορείτε να έχετε ένα αξιοπρεπέ εισόδημα μπορείτε να περάσετε στην επιχειρηματικότητα, αν δεν βρίσκετε δουλειά, και να βρείτε τέλο πάντων αξιοπρεπή εισόδημα. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινικό να το πει κανεί. Γιατί πολλέ φορέ αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Η επιχειρηματικότητα επουδενή δεν είναι το μέλλον. Γιατί υπονομεύει την αγορά εργασία και θα έχουμε μια παγκόσμια ανταλλαγή εργαζομένων όπου στην ουσία θα καταντήσετε να αναζητάτε δουλειά ή μεροκάματα των 10 λεπτών ή της ώρας. Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο συμφωνώ είναι το ότι αυτή η εργασία πλατφόρμας είναι ενδιαφέρουσα για και χρήσιμη σε φοιτητές και νοικοκυρές. Αν κάποιο έρχεται, α πούμε, κατάγεται από μια χώρα του κόλπου, ίσως να μην έχει πολλές δυνατότητες, αλλά στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, το να πούμε ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι καλές για φοιτητέ, νοικοκυρές και γυναίκες που που προέρχονται μάλλον κατάγονται από τις χώρες του κόλπου, αυτό θα πρέπει να το, να το δούμε κατά πόσο δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τελικά μια σωστή εργασία, μια σωστή μορφή εργασίας. Και τέλος, για τα δομένα. η Γιουνιρόπα μαζί με τη ΦΕΠΣ κάνουν κάποιες έρευνες εδώ και δύο χρόνια και έχουμε καλύψει, καλύψει αρκετές χώρες για αυτή την gig οικονομία. Είδαμε ότι μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού απασχολούνται σε αυτές τις νέες μορφές οικονομίας και έχει σημαντικό εισόδημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Καταρχάς να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Σούστερ και ζητώ συγγνώμη αν δεν ήμουν πολύ σαφή στην σύντομη παρουσίασή μου, ίσως να μην είχα αρκετό χρόνο. Για το θέμα των αυτοαπασχολημένων υπάρχει όντω ένα νομικό ζήτημα. Αλλά εγώ επικεντρώθηκα στου ε, αυτοαπασχολούμενου καταρχά για δύο λόγου. Για τα δεδομένα. Καταρχά, εμεί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι απασχολούμενοι βάσει των υπαρχόντων δεδομένων. Και επικεντρωνόμαστε στου αυτοαπασχολούμενου χωρί εργοδότε. Γιατί σε αυτέ τι περιπτώσει οι ίδιοι κατατάσσουν τον εαυτό του στου αυτοαπασχολούμενους όταν κάνουμε να τελειώσω αυτό καταρχάς και ο δεύτερος λόγος οποίους, για τον οποίο επικεντρώθηκα συγγνώμη στους αυτοαπασχολόμενους είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν την κατηγορία οικονομίας που συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι έχετε δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν νέα φαινόμενα, νέα δεδομένα που μεταβάλλονται γρήγορα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και το είπε και κάποιος άλλος για την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε τους κανόνες που διαθέτουμε ώστε να εντάξουμε τους ανθρώπους στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Και κάτι άλλο για τα δεδομένα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τρία πράγματα. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις πρόξεις μελέτε μας, μπορούμε να προσθέσουμε βέβαια ερωτήσεις για να βελτιώσουμε τη συλλογή των δεδομένων καμιά φορά χρειαζόμαστε και πιο ενισχυμένα δειγματολόγια, γιατί ίσω να είναι περισσότερος ο αριθμό, οπότε εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και επίση να περιλάβουμε διοικητικά δεδομένα, βελτιωμένα, αλλά και να ωφεληθούμε από την σύνδεση αυτών των ε, διοικητικών δεδομένων με τι έρευνε. Και τέλο θα ήθελα να πω ότι ο ιδιωτικό τομέα συλλέγει πάρα πολλέ πληροφορίε για αυτού του εργαζομένου. Οπότε χρειαζόμαστε ένα είδο ε, ΣΔΙΤ, όχι μόνο για φορολογικούς λόγους, αλλά για να υπάρχει σωστή ανταλλαγή αυτών των στοιχείων, αυτών των δεδομένων και συμβαίνει συχνά αυτή η ανταλλαγή, δημιουργώντας έτσι μια ροή πληροφοριών, ακολουθώντας βέβαια τη ροή του κεφαλαίου. Για τα δεδομένα επίσης να πω ότι επειδή γνωρίζουμε ελάχιστα και λένε διάφοροι ότι εντάξει υπάρχει ρευστότητα στην αγορά εργασία και μετακινήσεις αλλά στην ουσία δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Είχαμε ένα πρόγραμμα έρευνας του ΩΣΑ για να δούμε ακριβώς κατά πόσο αυξάνεται η κινητικότητα δηλαδή αν μπαινοβγαίνει ο κόσμος σε διάφορες θέσεις απασχόλησης. Αν δείτε τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, που έχουν στοιχεία αποδεικνύουν ότι έχουμε λιγότερη κινητικότητα από ό,τι σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει. Χρειαζόμαστε περισσότερε έρευνε και προσπαθούμε αυτό να το καλύψουμε στον ΩΣΑ. Για την επιχειρηματικότητα. Νομίζω πριν 10 χρόνια Μιλούσαμε για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας και είχαν δοθεί και κίνητρα για την προώθηση της αυτοπασχόληση και της επιχειρηματικότητας. Τώρα προσπαθούμε να τα αποσύρουμε κάποια από αυτά τα κίνητρα γιατί κατανοήσαμε ότι οδηγούν σε κάποιες τεχνητέ μορφές αυτοπασχόληση και εσφαλμένη κατάταξη στην αυτοπασχόληση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ένα Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών όπου μελέτησαν ακριβώς τις, ε, τα επιδόματα και τις φορολογικές εραφρύνσεις για τους απασχολουμένους. Αλλά αυτό το κάνανε για δικού του λόγου, επειδή ακριβώ είχαν ε, μορφέ συνταξιδότηση οι οποίε επεκτηνόταν και στου αυτοαπασχολούμενου και υπήρχαν κάποια γενά όσον αφορά τον ε, κρατικό προπολογισμό. Αλλά τέλο πάντων, σε σχέση με άλλα παραδείγματα από άλλε χώρε, για το τι κάνουν αυτές δηλαδή για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική πρόνοια. Είναι ευρύ ζήτημα αυτό και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις εισφορές, το πώς τακτικές είναι αυτές και το ενδεχόμενο να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις εισφορές. Στην Αυστρία ξέρω ότι υπάρχει ένας ατομικός λογαριασμός για κάθε απασχολούμενο, το οποίο σημαίνει ότι αν μετακινείσαι, αν μετακινείσαι δεν χάνεις δικαιώματα ε, που αφορούν αποζημιώσεις, ε, επιδόματα ανεργίας κλπ. Το ίδιο και στην Γαλλία διατηρείς το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας ακόμα και αν ε, βρεις δουλειά αν βρει μια εργασία ας πούμε, η οποία θα είναι μόνο εξάμηνη, δεν χάνει τα δικαιώματά σου για το επίδομα ανεργία. Οπότε αν είσαι πάλι άνεργο μετά από 6 μήνε, να συνεχίζει να τηρεί το δικαίωμά σου για επίδομα ανεργίας. Και τώρα για το κατά πόσο οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν μέσω των συσφορών τους να έχουν δικαίωμα σε συνταξιοδότηση, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά γιατί όντω εκεί υπάρχουν και κάποια κενά. Θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής ο κύριος Θεϊσακ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ερωτήσεις. Ένα ουσιαστικό ερώτημα είναι πράγματι τι είναι το όντω καινούριο και εδώ πέρα περνάμε στο θέμα της κατάταξης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είχαμε και πριν ε, τρίμερης ε, σχέσεις εργασίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η οικιακή βοηθή. Επίσης, ε, στην Ανατολική Ευρώπη κατά κανόνα μιλάμε για μικρο αυτοαπασχολούμενης. Πρέπει ακριβώς να δούμε το ότι γίνεται. Και Βεβαίω, ποιο είναι το σημαντικότερο θέμα, το θέμα της αποζημίωσης, το θέμα των αμοιβών. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να γίνουν 300 μελέτες όταν ο κόσμος ε, δουλεύει κανονικές ώρες πρέπει να αμείβεται με μια αμοιβή με την οποία μπορεί να ζει. Δεν είναι θέμα παραβίασης εδώ πέρα του ανταγωνισμού και νομίζω ότι είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό να πούμε ότι θα πρέπει να αμείβεται με μια χίτινη η εργασία. Και αυτό εντάξει σχετίζεται με την ε, τεχνολογία. Το νέο πλαίσιο είναι ακριβώς η τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία δεν είναι ένας μοιραίος αυτοματισμός. Εξαρτάται από εμά πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Χάρη Λέβερμαν. Έχει ε, γράψει διάφορα βιβλία για την υποβάθμιση της δουλειά στον 21ο αιώνα και περιγράφει ακριβώς ε, το φαινόμενο αυτό που αφορά την βιομηχανοποίηση της χειρονακτικής εργασίας. Και αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την βιομηχανική επαχή που περνάει στις υπηρεσίες γιατί μεταξύ μπορούμε να έχουμε τόσο μικρό μεμονωμένο έλεγχο σε άτομα. Δηλαδή, έχουμε πλέον πράγματα τα οποία παλιά μπορούσαν να γίνουν μόνο σε βιομηχανική κλίμακα. Π.χ. αυτός ο οποίος είναι trader ε, μετοχών. Αξιολογείται καθημερινά κάτι το οποίο γινόταν παλιά και για τον βιομηχανικό εργάτη. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και αυτό το οποίο είναι πραγματικά καινούριο είναι ακριβώς η εργασία στον ψηφιακό χώρο όπου υπάρχουν ακριβώς οι ε, νέες αυτές μορφές οι οποίες δεν είναι μόνο οι επισφαλείς. Μπορώ εγώ παραδείγματος χάρη να στείλω την δουλειά μου στην Ινδία, να την ελέγξει κάποιος και να μου την ξαναστείλει. Έχουμε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό με διαφορετικό όμως κόστος ε, εργασ... Ε, διαβίωσης εκεί που ζούμε. Αλλά δεν χρειάζεται από την άλλη πλευρά να στείλουμε, ξέρω την εργασία εκεί ή να φέρουμε το φθηνότερο εργαζόμενο εδώ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στον ψηφιακό χώρο και να μετατοπιστεί η εργασία. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι πού προσφεύγουμε, πού μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε εμεί μια σύμβαση εργασίας, ξέρω εγώ, που να είναι σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, τι ε, ισχύ έχει όταν ο εργοδότης μου είναι Ινδός ή Αμερικανός παραδείγματο χάρη. Ναι, έχουμε διαφορετικά νέα προβλήματα και βεβαίως έχουμε και το θέμα το ότι ε, ρυθμίζαμε τις τιμές των αυτοαποσχολούμενων Μα αυτό γινόταν επί αιώνες. Δεν... Τον 19ο αιώνα είχαμε πλήρη ανταγωνισμό και εκεί πέρα ακριβώς ανεπτύχθηκαν τα συνδικάτα οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις, πράγματα τα οποία έχει δεχτεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαμε κάποιες συγκεκριμένες εξαιρεσει από το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Λέμε, χρειαζόμαστε κοινωνικούς εταίρους, ε, επικουρικότητα κτλ. Λοιπόν, και λέμε δεν έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ε, για αυτές τις ε, μονάδες. και πρέπει να δούμε ακριβώς ε, με ποιους ε, διαπραγματευόμαστε με τους καταναλωτές ε, ή με κάποιον άλλον. Και βεβαίω έχουμε το θέμα της μεταβολής των αξιών. Και το βασικό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι και τα άτομα αυτά, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους διαφορετικά και θεωρούν ότι είναι ανεξάρτητοι, δεν αναζητούν αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, αλλά περισσότερο ανταγωνισμό. Και τι σημαίνει ο ανταγωνισμός? Στην τιμή. Και το θέμα είναι ακριβώς ε, σε ποιο βαθμό θα φτάσει αυτός ο ανταγωνισμός στην τιμή. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ όλους τους ειδικούς μας. Νομίζω ε, είμαστε και σε, θα είμαστε και σε στενή επαφή. Καλώς ορίζω και την εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και παρακαλώ για το σχόλιο σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μαρία Νιμπέρ, Γενική Διεύθυνση Έμπλ, από την Διεύθυνση Δεξιοτήτων. Συνερπαστική συζήτηση, πραγματικά. Συνερπαστικές οι παρουσιάσεις. Δύο λόγια το ψήφισμα για την συμμετοχική οικονομία, την συνεργατική οικονομία. Ετοιμάζουμε σχόλια. Όσον αφορά τα στοιχεία όμω και την πρόσβαση στα δεδομένα, το τονίζουμε αυτό ως θέμα στο θεματολόγιο ήδη από πέρσι. Ε, τονίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων, έλλειψη πληροφοριών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι μας αφορά, για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό. Συνεργαζόμαστε με την Eurostat, για να βελτιώσουμε τη θέση μας και μελετούμε και παρακολουθούμε μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν πολλές από αυτές στη δική μας Γενική Διεύθυνση για να κατανοήσουμε καλύτερα εν τέλει τον αντίκτυπο στην οικονομία των συνεργατικών μορφών δραστηρι... οικονομικής δραστηριότητας. Πολύ ενδιαφέρον το χείριμα. Περιμένουμε πληρέστερα στοιχεία του χρόνου, δεύτερο τρίμηνο και εννοείται θα σας ενημερώσουμε. Συζητούμε επίσης θέματα δήλωτης εργασίας, σε πλατφόρμες έχουμε την Επιτροπή Διαλόγου για την προσωρινή εργασία. Εξετάζουμε τον γενικότερο οικονομικό αντίκτυπο, όπως είπα, της εργατικής οικονομίας. Μία ομάδα στοιχείων που είναι ενδιαφέροντα, θεωρώ, εν προκειμένου είναι το εξή. Η, Καναδική Στατιστική Υπηρεσία πριν από μερικέ μήνε εξέδωσε μελέτη, στο πλαίσιο τη οποία εξετάζουν και τι πλατφόρμες α πούμε στον τομέα των μεταφορών ή τη στέγη τη της κατοικίας, μεταξύ καταναλωτών. Η ανταλλαγή υπηρεσιών δηλαδή μεταξύ καταναλωτών. Εκεί διαπιστώνουμε ότι μόνο 1%, λιγότερο μάλιστα, 1 του 1% των εργαζομένων σε αυτού του τομεί είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Λιγότερο από 1%. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, ω ε, στατιστικό έβριμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω όλα. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις μόνο. Πρώτη παρατήρηση. Αυτά τα οποία είπε ο Χάιντς Μπέκερ για κοινωνική οικονομία της αγοράς και όχι ελεύθερη ε, αγορά. Ε, να σας υπενθυμίσω, το υπενθυμίζουμε και εδώ. Κοινωνική οικονομία της αγοράς σημαίνει ότι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται. Βλέπουμε εδώ πέρα τις συγκλονιστικότερες ε, εξελίξεις τα τελευταία 100 χρόνια στον κόσμο της εργασίας. Αν ε, όχι και σε περισσότερες ε, σε, σε μεγαλύτερο βάθος Λοιπόν, ο καθηγητής ανέφερε και τη Λευκή Βίβλο της Γερμανικής Κυβέρνησης για την εργασία 4,0 όπως λέγεται και μιλάμε εκεί για μεγάλες ανατροπές που απαιτούν κάποια κοινωνική ρύθμιση. Αφενός λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει εδώ πέρα να δραστηριοποιηθούν, αλλά πολλά πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να ρυθμιστούν και από την κοινωνία, από την πολιτική, όχι στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά λόγω του ε, διασυνοριακού χαρακτήρα αυτών των ε, μορφών εργασία ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, να το πιέμε, για να ρωτιόμουν τις τελευταίες εβδομάδες από μακριά βλέποντας ε, τα θέματα αυτά ε, από το κρεβάτι του νοσοκομείου για τα κοινωνικά δικαιώματα πουθενά εκεί πέρα δεν υπήρχε κάποια σύνδεση στον κόσμο των ΜΜΕ, όχι το τι ακούγεται εδώ μέσα, αλλά ακόμα και για ανθρώπους που είναι μέσα στο σύστημα όπως εγώ, στη δημοσιότητα το θέμα λοιπόν ήταν ένας ευρωπαϊκός πυλώνας ε, κοινωνικών δικαιωμάτων ή όχι, δεν έπαιζε κανέναν ρόλο. Δηλαδή έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ως βουλευτές για να θέσουμε το θέμα. Και... Βεβαίω ε, να έχουμε κοινωνικά δικαιώματα τα οποία δεν θα είναι απλά μια χειρονομία αλλά θα μπορεί ο κόσμος έτσι να διασφαλίζει την ε, διαβίωσή του το οποίο πρέπει να κάνουμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Είναι θα πρέπει να εμποδίσουμε την επανεμφάνιση ε, ξανά του ούτε καν του μεροκάμα του, του, της δουλειάς αυτής με την ώρα. Ε, μιλάμε καν για για μεροκάματο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση. Ευχαριστώ τους ειδικού, ευχαριστώ την Κομισιόν. Οπωσδήποτε το θέμα θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε ακόμα 8 λεπτά μέχρι να ξεκινήσουμε. Οπότε οι τεχνικοί μας ε, που ασχολούνται με το θέμα μπορούν να ξαναξεκινήσουν να κάνουν ε, θόρυβο και εμείς θα κάνουμε 8 λεπτά διάλειμμα.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 Can you hear me? Okay, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 Έχουμε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες εδώ. Βοηθούν πάρα πολύ όταν έχουμε άτομα με αναπηρία. Και ερχόμαστε εδώ λοιπόν για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Η συγκίτρια είναι η Χέλγκα Στίβενς. Τη διαδικασία την ξέρετε νομίζω. Μπορούμε σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε την μετάδοση του κειμένου. Έχουμε και τις κόκκινες ε, και κίτρινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο μιλητής. Η κίτρινη κάρτα είναι για να πείτε ότι μιλάει πολύ γρήγορα ομιλητής και πράσινη κάρτα είναι ότι όλα πάνε καλά. Αυτά. Λοιπόν, ε, θα τα αφήσουμε όμως, μην πάρετε τις κάρτες μαζί. Οπότε, περνάμε τώρα στο θέμα αυτό. Έχουμε τέσσερις ε, πάλι εμπειρογνώμονες. Ε, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης εδώ πέρα ε, είναι αρμόδια. Έχουμε την Άντια Χαντάτ από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, τη Ροζίτα Χίκη από το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και η Τάνια Τάτζιτς, αντιπρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ με βίντεο Αυτό ήταν ο θόρυβο που ακουγόταν γιατί ο τεχνικός εκεί προσπαθούσε να δημιουργήσει μία σύνδεση. Για να μπορέσουμε ακριβώς ε, να ακούσουμε την κυρία Τάτζιτς. Λοιπόν, τον λόγο έχει ο Μανουέλ Τράουνς από τη Γενική Διεύθυνση Αποσχόλησης πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση προς την Κομισιόν να παρουσιάσει την έκθεση υλοποίηση της στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως την κυρία Στίβενς ε, για το έργο της, πολύ χρήσιμο για το μέλλον, για την ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά και για τη συνεχεία της πολύ γρήγορα η στρατηγική εγκρίθηκε για να επιτρέψει την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αναπήρων. Και για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά με την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά κυρίως την προσβασιμότητα, την συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση. Η έκθεση που εγκρίναμε τον Φεβρουάριο του 2017 είναι έγγραφο εργασίας, ένα εσωτερικό έγγραφο της, ε, των υπηρεσιών της Κομισιόν που δεν αποτελεί αξιολόγηση, δεν αποτελεί επίσημη αξιολόγηση. Αυτό θα το κάνουμε στο τέλος της περίοδου τη της στρατηγικής. Ή να θέλετε μια ματιά στο μέλλον, καταγράφει τα όσα μένει να γίνουν και καταγράφει βεβαίω και αυτά τα οποία ήδη έγιναν στο πλαίσιο της υλοποίηση της στρατηγικής. Τι κάναμε λοιπόν και τι μένει να κάνουμε σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα. Ομολογώ ότι θέλαμε να είμαστε έτοιμοι πιο νωρί, όμως α, μεσολάβησε ένας πολύ επικοδομητικός δημόσιος διάλογος με σειρά ακροάσεων που κατέληξε σε πάνω από 1.600 απαντήσεις. Η ανάλυση πήρε λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μάλιστα θα το βρείτε σε ένα από τα παραρτήματα της έκθεσης, όπου αντικατοπτρίζονται οι βασικές ανησυχίες, τα βασικά μελήματα, αν θέλετε, όπως προέκυψαν από αυτήν την διαβούλευση, κυρίως για τα θέματα απασχόλησης των αναπήρων. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα στην έκθεση, αλλά το πρώτο που προέκυψε το πιο σημαντικό είναι αυτό. Στο παράδειγμα της έκθεσης θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα, το οποίο επισέρχονται σε περισσότερες λεπτομέρειες διαφορών πτυχών της στρατηγικής, βάσει και των ε, συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το παράδειγμα 5 είναι πολύ χρήσιμο, διότι καταγράφει αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα νομοθετήματα των τελευταίων ετών στο πλαίσιο και της στρατηγικής, όλα επίκαιρα και τα οποία συνδέονται με την αναπηρία. Δεν είναι λεπτομερής καταγραφή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ή της Ένωσης γενικότερα σε θέματα αναπηρίας. Αυτό ε, θα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο και πρέπει να εγκριθεί και επισήμω. Όμως, είναι δουλειά που πήγε σε αρκετό βάθος, καταγράφει, όπω είπα, διάφορα νομοθετήματα και τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία. Όπως ε, προείπα, μαζέψαμε 130 τέτοια κείμενα, τα οποία διαπώνουν την ευρωπαϊκή δράση. Ως προς τα συμπεράσματα αυτού του εγγράφου εργασία. Φαίνεται ότι ο γενικός στόχος της στρατηγικής παραμένει πάντοτε επίκαιρος παρά την πρόοδο. Φαίνεται ότι κάναμε σωστές επιλογές ως προς τους στόχους, όμως πρέπει να συνεχίσουμε ως το τέλος της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, δηλαδή το 2020. Και δει στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης. Δεν χρειάζεται να πω ότι η Κομισιόν παραμένει προσιλωμένη στον στόχο του 2020. Να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων που υλοποιήθηκαν. Εγκρίναμε πρόταση, για παράδειγμα, την European Accessibility Act, την, πράξη, την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, μία άλλη για τους ιστοτόπους, μία άλλη για τις μεταφορές, και πάλι θέματα πρόσβασης και βοήθειας προς άτομα με αναπηρίες. Μια άλλη πιλωτική δράση σε οκτώ κράτη-μέλη. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αλλά την τρέχουν 8 κρατημέλη. Επίση, έχει γίνει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων. Διότι η κατάρριξη των διακρίσεων και η προσβασιμότητα ε, είναι στοιχεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, πρόδωσε διάφορους δείκτες, το έρασμος, το έρασμος το οποίο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. Έγινε πολλή δουλειά λοιπόν που εν γέννη κρίνεται θεωρώ θετικά. Πρόκειται για καταγραφή βεβαίω για μια πρώτη καταγραφή πεπραγμένων. Δεν πέντε την Κομισιόν για τα όσα έκανε, απλώς καταγράφουμε όπως είπα. Από εδώ και πέρα όμω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά, μετά την περίοδο 10-20. Το έγγραφο εργασία δεν λέει κάτι σχετικά. Είναι προφανώ όμω ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την επίσημη αξιολόγηση τη στρατηγική, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε μετά το 20. Το ερώτημα κλειδί είναι, χρειαζόμαστε, συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία. Ε, με ποια μορφή, ποια διάρκεια, σε ποιου τομεί, σε ποιου κλάδου κλπ. Είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα αυτά. Θα δούμε τι θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου συζητήσεων από την κυρία Στίβενς. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Από εκεί πέρα εσείς ε, μπορείτε να συνεχίστε πάνω στον δρόμο που άνοιξε το έγγραφο εργασία. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον διάλογο αυτόν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η Νάντια Χαντάτ από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας για 7 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσετε σε αυτόν τον διάλογο. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Περαμένει των δικαιωμάτων 18 εκατομμυρίων αναπήρων στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή ΕΜΠΛ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Στίβενς, συμμετέχουν στον διάλογο λαμβάνοντας υπόψη το 4.2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Ευχαριστούμε που από την αρχή της συζήτησης καλέσετε και αναπήρους και εκπροσώπους αναπήρων. Από αυτήν την έννοια ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στον διάλογο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστηρίζουμε την κυρία Στίβενς και την Επιτροπή στο πλαίσιο και στη διάρκεια εκπόνησης της σχετικής έκθεσης. Για μας, τα βασικά σημεία που πρέπει να τονίσουμε είναι τα εξή. Η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση μέτρων, στο πλαίσιο της υλοποίησης δηλαδή των ε, δράσεων που υποστηρίζει και το φόρουμ μας. Είναι επίσης ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς ένα κείμενο του 2015, αξιολόγηση υλοποίησης ε, μέτρων, Κάτι το οποίο πρέπει να διαβάσουμε σε συνάρτηση και με την έκθεση αξιολόγηση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί και επαναδιαμορφωθεί εκ βάθρων για τα επόμενα χρόνια, 17 έως 20. Καλούμε επίσης τη συνέχιση των προσπαθειών για την υλοποίηση τη στρατηγική και τη διαμόρφωση μια νέα για την περίοδο 2020-2030, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι πτυχέ τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει σε πρώτη φάση βεβαίως να αξιολογήσουμε την κατάσταση, των δικαιωμάτων των αναπήρων και να τα αξιοποιήσουμε αυτά διαμορφώνοντας τη νέα στρατηγική. Να προσθέσουμε νέους τομείς, νέες πτυχές, τα οποία όπως προείπα θα τα συνδέσουμε με την αναθεώρηση διαφόρων άλλων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, να ρηθούν αυτά υπόψη στην πολιτική ισότητα ε, των δικαιωμάτων των παιδιών και στην εξωτερική δράση. Αυτά βάσει ενό σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης με διαμέσους στόχους και δείκτες. Διότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία υιοθετήθηκε πριν από την CRPD στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς η επόμενη στρατηγική πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εφαρμογή της CRPD. Η στρατηγική λοιπόν για το 2020-2030 πρέπει να συμπεριλάβει και να εμπλέξει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλους τους οργανισμούς της, και να λάβει υπόψη τα συμπεράσματά μας για το μέλλον. Η στρατηγική πρέπει να είναι πλήρως ενταγμένη και συνδεδεμένη με τις κοινωνικές και μακροοικονομικές πολιτικές. Την πολιτική επίσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ούτω καθεξής. Η στρατηγική πρέπει επίσης να ενσωματώνει τους στόχους αηφορίας και τους στόχους της στρατηγικής των ΗΕ ΕΕ για την περίοδο 2020-2030. Συνεπώς, το 2021 πρέπει να κηρυχθεί το νέο έτος για τους αναπήρους. Να συνεχίσουμε λοιπόν τον διάλογο. Να συνεχίσουμε να τονίζουμε τα βασικά θέματα, τα βασικά προβλήματα που θέλουμε να ληφθούν υπόψη ως θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος, πώς λέμε, και που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής για τους αναπήρους. Για να σωματωθεί λοιπόν η προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων σε όλες τις πολιτικές, χρειαζόμαστε μια οριζόντια, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί οι νόμοι, οι πολιτικές, τα προγράμματα πρέπει να εναρμονιστούν με την CRPD. Πρέπει οι ανάπηροι εν τέλει να συμμετάσχουν οι ίδιοι στη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος. Καλή λοιπόν η καταγραφή, αλλά πρέπει να καταγράψουμε και τους τομείς στους οποίους υστερούμε, να δούμε πού υστερούμε, πού υπάρχουν λήψεις στην νομοθεσία, στην νομοθετική διαδικασία, στην ασωμάτωση στην απείρια στις άλλες πολιτικές και στην υλοποίηση της CRPD. Αυτά πρέπει να κάνουμε και ειδικά η καταγραφή των ελλείψεων πρέπει ρητός να συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία. Η CRPD προβλέπει επίση την συμμετοχή και την εκπροσώπηση των αναπήρων στην διαδικασία της υλοποίηση και τη εφαρμογή τη σύμβαση. Η επόμενη φάση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής πρέπει να υλοποιηθεί μέσω δομημένου ευέλικτου διαλόγου όχι μόνο με τους διάφορους οργανισμούς αλλά και με το κίνημα των αναπήρων. Στο άρθρο 4.3 και 4.5 της ΕΠΔ ΕΕ αυτά προβλέπονται ρητός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πρέπει να θεσπίσει ένα πρόγραμμα για τους τους οργανισμούς εκπροσωπή των αναπήρων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν την εντολή του. Και τέλος, συστήνουμε διαθεσμικό συντονισμό ε, και μάλιστα τη δημιουργία ενό σχετικού μηχανισμού, ο οποίος θα διευκολύνει το παρέσμα στην εποχή και την ομαλή υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία. Περαιτέρω την υλοποίηση της Σύμβασης των Εθνών και τη συμμετοχή των αναπήρων σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ακολουθεί η Ροζίτα Χέκε από το γραφείο του Διαμεσολαβητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κυρίε ε, και κύριοι, κυρία Στίβεν, σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε. Σήμερα εκπροσωπούμε το πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία και την σχετική σύμβαση που προωθεί και επιτηρεί την ε, εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από το Κοινοβούλιο, το Γραφείο του Δημοσιολογητή, την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, ε, το οποίο μόλις ακούσαμε. Και Όλα τα μέλη έχουν συνεισφέρει για να μπορέσουμε ακριβώς να δούμε ποια είναι τα καθήκοντα και η εντολή που έχουμε. Πριν ε, σχολιάσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρία, θα ήθελα να αναφέρω δύο πρόσφατες δραστηριότητες του πλαισίου που νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι βουλευτές. Τον Απρίλιο του 2017 συναντηθήκαμε με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα ενσωματωθεί η πολιτική της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξωτερική δράση, στις δηλώσεις αρμοδιότητας της Ένωσης και στην δυνατότητα να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει ατομικές προσφυγές ενώπιον της σχετικής επιτροπής. Και τον Μάιο του 2017 είχαμε την τέταρτη ετήσια συνάντησή μας με τα εθνικά πλαίσια για να ανταλλάξουμε ορθές πρακτικές για την παρακολούθηση της σύμβασης. Εστιαστήκαμε στο άρθρο 19 της σύμβασης στο δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης και συγκεκριμένα στην χρήση διαρθρωτικών και επενδυτικών κονδυλίων για να το στηρίξουμε αυτό. Οπότε αυτές οι κοινέ δραστηριότητες προφανώς συμπληρώνουν το έργο των μεμονωμένων μελών του πλαισίου για να προωθήσουμε και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της σύμβασης. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία, όπως ξέρουμε, η στρατηγική είναι το κύριο μέσο για να στηρίξουμε την εφαρμογή της σύμβασης από την Ένωση και γι' αυτό το λόγο η αναθεώρηση αυτή και η εκδήλωση σημερινή έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως ξέρουμε από την έκθεση της Κομισιόν έχουμε επιτύχει πρόοδο περιλαμβανομένης της ε, οδηγίας για προσβασιμότητα του δικτύου και την ευρωπαϊκή πράξη περί προσβασιμότητας. Επίσης, σε οτιδήποτε χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα προσβασιμότητας, αλλά και αιρεσιμότητα εξ ante όταν θα περάσουμε παραδείγματο χάρη από την θεσμική φροντίδα σε φροντίδα εντό της κοινότητα. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να αναλάβει δράση και σε άλλου τομείς περιλαμβανομένη ε, και τη οδηγία ίση μεταχείρισης. Η σχετική επιτροπή στον ΟΗΕ στην Γενέβη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταρτήσει ξεκάθαρες κατευθυντήριες ε, γραμμές για να περιληφθούν δείκτες ε, και ξεκάθαρα μέτρα σύγκρισης για το εάν περιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν τον Ιούλιο του 2016 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν ε, επί τη ευκαιρία της αναθεώρησης της στρατηγικής να περιλάβει και την διάσταση του φίλου και στις δεσμεύσεις της εξωτερικής δράσης με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και πάλι με συγκεκριμένους δείκτες μετρήσιμους. Πέρα από το ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου το πώς ε, εφαρμόζονται στην πράξη τα της παρακολούθησης και έτσι διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα. Πρέπει να εστιάζουμε στις ε, υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, το πώς επηρεάζει η λιτότητα τα άτομα με αλλά και την ε, κατάσταση με τους πρόσφυγες, για να αναφέρω δύο επίκαιρα παραδείγματα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τα μέλη του πλαισίου, συμμετείχαμε στην δημόσια διαβούλευση για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής αυτής. Επίσης επισημάναμε ότι η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα έτσι ώστε οι καταληκτικές παρατηρήσεις της σχετικής επιτροπής, παραδείγματο χάρη για την χρήση των διαρθρωτικών κοντιλίων, θα εφαρμοστούν. Νομίζω πως είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι οργανώσεις αυτές ε, ζήτησαν και την πολιτική ε, συμμετοχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Παραδείγματο χάρη πρότεινε η η Υπηρεσία των Δικαιωμάτων να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα, κυρίως μέσω κατευθυντήριων γραμμών για τα δημόσια κτίρια. Το φόρουμ της προσβασιμότητας είπε πως η άρνηση των δικαιωμάτων με κοινωνικο-ψυχολογικές δυνατότητες ε, από το να ψηφίζουν τους αφαιρεί δικαιώματα. μπορούσαμε έτσι να βοηθήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα μέτρα μέσω συμβουλευτικών φορέων που θα περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. Επίσης θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τις ευκαιρίες για συμμετοχή στην διαβούλευση μέσω της ευρύτερης δημοσιότητας, μέσω οδών που είναι πιο προσβάσιμες. Επίσης ετέθη το, το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών με αναπηρία. Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα του τι έχουμε κάνει. Για το μέλλον θα έλεγα ότι απαιτείται μια νέα ολιστική στρατηγική χωρίς την οποία δεν θα εφαρμόσουμε σωστά την σύμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ περνάμε τώρα στον τέταρτο εμπειρογνώμονα να δούμε τι θα γίνει. Καλωσορίζω την κυρία Τάντζιτς, αντιπρόεδρο της σχετικής επιτροπής για την σύμβαση με Skype από το Βελιγράδι, αν έχω καταλάβει καλά. Λοιπόν, έχετε τον λόγο για 7 λεπτά. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, βουλευτές του Κοινοβουλίου, συνάδελφοι, ελπίζω να με ακούτε καθαρά και δυνατά να ευχαριστήσω και τους τεχνικούς για τη θαυμάσια υποστήριξη. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να είμαι εκεί διαζώσεις, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσα να σημειώσω αυτό το σημαντικό ζήτημα. Να ευχαριστήσω και την κυρία Στίβενς για την ευγενή της πρόσκληση να σας μιλήσω σήμερα. Πριν από δύο χρόνια και παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιασε την πρώτη της αρχική της έκθεση στην Επιτροπή. Ένα ιστορικό γεγονός για πρώτη φορά ένας περιφερειακός οργανισμός ο οποίος συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και που είναι μέρος αυτής της σύμβασης των δικαιωμάτων παρουσίαζε ένα τέτοιο έγγραφο. για τις συστάσεις της Επιτροπής. Μια από, αυτή, μια από αυτές ήταν η ταχεία υιοθέτηση της νομοθεσίας που αφορά την πρόσβαση. Να ευχαριστήσω λοιπόν το Κοινοβούλιο και το ρόλο που διαδραμάτισε. Παρ' αυτά Μας ακούτε παρακαλώ στην αίθουσα. Μας ακούτε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για την περίοδο 2017 με 2020 να υπάρχει μια ξεκάθαρη εφαρμογή των συστάσεων του σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και ελπίζω πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική ε, προσεχώς και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια στρατηγική μετά το 2020 η οποία πραγματικά θα βασίζεται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων ε, με Αναπηρία. Οπότε, αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας ε, και ελπίζω να ακούστηκα καλά. Και μας συγχωρείτε, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με την ε, διερμηνία. Και βεβαίως είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και αναμένω και τις ε, περαιτέρω ερωτήσεις και συνεργασία. Das waren die vier Experten. Σας ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι τέσσερις ειδικοί μας. Παίρναμε συζήτηση τώρα. Τον λόγο έχει η κυρία Χέλγα Στίβενς. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Colleagues. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, εμπειρογνώμονες, καταρχάς να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που μίλησαν εδώ σε αυτή την συζήτησή μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία σας που διασφάλισε την εξαγωγή αυτής της συνάντησης που ήταν τόσο σημαντική σε σχέση με την συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και εκπροσώπων τους. Εγώ ιδιαίτερα χαιρετίζω την βούληση της Κομισιόν για την συνεργασία με το Κοινοβούλιο για την στρατηγική αυτή και πέραν του 2020. Θα ήθελα να τονίσω ότι το σχέδιο εκθεσής όπως θα κατατεθεί αυτή τη βδομάδα είχε συνταχθεί σε στενή συνεργασία με το EDF, τα μέλη του και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εργάζονται πάνω σε θέματα ισότητας και εξέλιξης διακρίσεων. Πριν από λίγες εβδομάδες μετά τη τελευταία συνάντηση το γραφείο μου είχε 8 workshop, 8 εργαστήρια διαλόγου για αυτά τα θέματα που κατέληξαν σε πολύ χρήσιμες παραγράφους ε, σε σχέση με το σχέδιο της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να επαφοηθώ τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Άνταμ και τη Μάριον τους αδέλφους που μίλησαν στα workshops, στα εργαστήρια αυτά και να ευχαριστήσω και όσους έστειλαν εκπροσώπους. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την ευκαιρία. Νομίζω ότι στάθηκε το σχέδιο έκθεσης στο EDF και στα μέλη του ώστε να διασφαλίσουν το ότι όλα τα σχόλια που θα κατατεθούν θα ενσωματωθούν με το σωστό τρόπο. Παράλληλα, συνεργάστηκα με το ETF και τα μέλη του για διάφορες τροπολογίες. Επειδή βέβαια το αρχικό μέγεθος της έκθεσης περιορίζεται σε κάποιες μόνο συγκεκριμένες σελίδες. Μέσω των τροπολογιών, εγώ θα προσπαθήσω να διασφαλίσω το ότι θα ληφθούν υπόψη όλα τα σχόλια. Το γραφείο μου θα στείλει τις τροπολογίες για υπογραφή σε όλους τους σκιώδες εισηγητής και άλλους αρμόδιους ε, ευρωβουλευτές πριν από την προθεσμία της 6ης ε, Σεπτεμβρίου ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος. Βεβαίως έχουμε τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά παρόλα αυτά περισσεύει χρόνος. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε πρόθεση να καταθέσετε τροπολογίες, ε, πείτε το στους συνεργάτες μου. Και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας, μαζί με τις οργανώσεις και τους συναδέλφους τους ε, συνεισηγητές και αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή απορία σε σχέση με την ε, έκθεση της τροπολογίας, σας παρακαλώ να έρχετε σε επαφή μαζί μας. Και ευχαριστώ επί τη ευκαιρία και τους ε, εισηγητές σήμερα, γιατί οι εισηγήσεις τους αποδείχθηκαν πάρα πολύ χρήσιμες και σας ευχαριστώ όλους πραγματικά που επιτρέψατε να γίνει αυτή η δουλειά και τη διευκολύνατε και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ κόσμος. Ακούσουμε τώρα τη συνάδελφα από το ΕΛΚ. Συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που λαμβάνει η χώρα αυτή η συνάντηση. Ελπίζω οι καρποί αυτής της συζήτησης να αποτελέσουν την τελική έκθεση για αυτή τη στρατηγική. Ως σχεδόν εισηγητής ήρθα σε επαφή με διάφορους ενδιαφερόμενους σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και τις προσδοκίες τους σε σχέση με το μέλλον. Απέστειλα ερωτηματολόγια σε ενδιαφερόμενους, διοργανώσαμε εργαστήρια ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στην ε, σύνταξη της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα σύντομα να σας μιλήσω για κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια των εργαστηρίων. Καταρχάς, οι συμμετέχοντες εκεί τόνισαν την ανάγκη για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όσον αφορά την ύπαρξη αυτής της ίδιας της στρατηγικής και μια εκστρατεία προώθησης και ενημέρωση θα ήταν πολύ καλή. Επίσης, οι συμμετέχοντες τόνισαν το ότι θα πρέπει να υπάρξει για τη στρατηγική αυτή ιδιοποίηση, ανάληψη της δηλαδή και πρόθεσή της. Θα πρέπει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο ενεργή στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, γιατί πιστεύουμε ότι οι μέθοδοι και τα μέσα σύγχρονης επικοινωνίας, όπως επίσης και η συμμετοχή των εθνικών αρχών αλλά και τη Κομισιόν θα μπορούσαν πραγματικά να επιτρέψουν την υλοποίηση αυτή τη στρατηγική. Νομίζω ότι με αυτή τη συνεργασία και με αυτή την επικοινωνική στρατηγική θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, πολύ καλύτερα δηλαδή από ότι αν περιοριζόμασταν σε μια διαδικασία διαβούλευση στην ιστοσελίδα τη Κομισιόν. Νομίζω ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εμπλακούν και να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της στρατηγικής αυτής, δηλαδή από τη χάραξή της, στον προγραμματισμό, μέχρι την εφαρμογή της και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η περίοδος από το 2020 μέχρι το 2030, γιατί υπάρχουν ανησυχίες και ερωτηματικά σε σχέση με το πώς θα αναθεωρηθεί ή θα αξιολογηθεί αυτή η στρατηγική και πώς θα μπορούσε να συνδεθεί βεβαίως με άλλες νομοθεσίες όπως η νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση ή την προσβασιμότητα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι θα θέλαμε η στρατηγική να κάνει περισσότερες προβλέψεις πρόνοιες σε σχέση με την ύπαρξη συστημάτων αρρωγής για όσους μένουν μόνοι τους επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις μεμονωμένες οι οποίες αφορούν αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και το ζήτημα της ε, εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας παρακαλέσω να τηρήσετε όμως τα δύο λεπτά. Μαρίτα Ούλφσκοκ κατόπιν ε, εκπροσωπεί την Ηλία Μπλινκεβίτσι ούτε ευχαριστώ. Τα βασικά σημεία της ομάδας μας εδώ είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην στρατηγική για να εφαρμοστεί η σχετική σύμβαση. Πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει μια σωστή δομή παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η στρατηγική δεν λαμβάνει υπόψη τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στα δικαιώματα τόπων με αναπηρία. Ξέρουμε ότι τα άτομα με αναπηρία βασίζονται στην κοινωνική προστασία και ξέρουμε πόσο ευπαθή είναι στην αγορά εργασίας και είναι πραγματικά αυτό ένα θέμα το οποίο επηρεάζεται από την οικονομία. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της ε, οικονομικής κρίσης ε, στα άτομα με αναπηρία για να κάνουμε κάτι. Και τρίτον, έχει μεγάλη σημασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρία του 2020 και 30. Δύο χρόνια έχουν απομείνει πριν ε, εκπνεύσει η τρέχουσα στρατηγική και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη περίοδο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να σέβεται τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με αυτήν την σύμβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ Μαριάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση σήμερα το πρωί που θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη. Αχα, κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τους εισηγητές. Ποιες είναι οι δράσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα που θεωρείτε ότι τηρούν αυτά που προβλέπει το CRPD Ξέρω ότι υπάρχουν τα θέματα προσβασιμότητα, κάποια άλλη αναφέρθηκαν σε άλλε δράσεις, αλλά θα ήθελα να μάθω το τι πήγε καλά και τι πήγε λιγότερο καλά όσον αφορά ας πούμε, θέματα νομοθεσίας ή κατευθυντήριο γραμμών. ή αν κάτι το οποίο προϋπήρχε δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι μαθήματα μπορούμε να αποκομίσουμε. Επίσης, θα ήθελα να μάθω συγκεκριμένα Ποιε δράσεις χρειαζόμαστε στη νέα στρατηγική για την αναπηρία, για την εφαρμογή του ΣΥΑΠΗΤΗ. Ακούσαμε, ας πούμε, για το mainstreaming, την ένταξη αυτών των πολιτικών στις υπόλοιπες πολιτικές, θέματα όπως ε, συμμετοχή των ατόμων κτλ. Αυτά θεωρώ δεδομένα, αλλά ίσως συγκεκριμένα και ιδιαίτερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τα θέματα προσβασιμότητας που το ανέφερε ο κ. Υπάρχουν άλλοι τομείς ή άλλες περιπτώσεις όπου για να εφαρμοστεί το ECRPD πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα πέραν της προσβασιμότητας που βεβαίως την συζητήσαμε διόντως σήμερα το πρωί. Θα θέλω να ακούσω τις απόψεις σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα η Τατιάνα Σντάνοκα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Χέλκα Στίβεντς και τη Γραμματεία για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης σήμερα. Μαζί με διαφορές ΜΚΟ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Βεβαίως αναμένουμε το έγγραφο ώστε να καταθέσουμε τροπολογίες. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ευρία συνένεση για το ότι θέλουμε να πετύχουμε και με βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να συνυπογράψουμε τις τροπολογίες που είπε η Χέλγα ότι θα καταθέσουν από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες. Τώρα για τη δομή της έκθεσης Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τους τομείς προτεραιοτήτων, αλλά και επιπλέον τομείς για δράσεις, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρίες. Επίσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης, το πιο σημαντικό κομμάτι της έκθεσης νομίζω ότι πραγματικά θα είναι αυτό που αφορά το μέλλον, δηλαδή στρατηγική μέχρι το 2030. Οπότε τις ευχές μου προς την Χέλγα και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε σωστά. Ευχαριστώ η κυρία Κούνεβα τώρα για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ευχαριστώ με την Επιτροπή και τους ειδικούς για τις πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις τους που βοηθούν. Αλλά έχω την αίσθηση πως βρισκόμαστε μόνο στο ξεκίνημα μιας τεράστιας δουλειάς που πρέπει να γίνει. Μιας δουλειάς η οποία να περιλαμβάνει μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε για την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά παράλληλα και με προτεραιότητα μέτρα για την ορατότητα του προβλήματος. Συνητήσω να λέω πως όσο λιγότερα γνωρίζει η κοινωνία για μας και τις δυσκολίες μας, τόσο χειρότερες αποφάσεις τα λαμβάνονται για μας χωρίς εμάς. Χαίρομαι για την δουλειά που έκανε η συνάδελφος και η συγκίτρια της έκθεσής μας, Χέλγα Στίβανς, με την ανταλλαγή απόψεων με τους επιρρογνώμοντες τους τομείς προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αναπηρίας. Χρειαζόμαστε ανάλυση των πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί, συγκεκριμένες πληροφορίες για την επιτυχία ή την αποτυχία τους και τους λόγους που δεν αποδείχτηκαν ως αποτελεσματικές ελπίζαμε. Χρειαζόμαστε πιο γρήγορο βήμα για ό,τι δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και πάλι τους λόγους για τους οποίους είχαμε μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε και προσεκτικότερο σχεδιασμό για το μέλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις καταπληκτικές δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Πρέπει επίσης να είναι σαφές πως τα προβλήματα μας είναι προβλήματα προτεραιότητες και για ποιο λόγο. Σκληρά χωρίς γνώσεις, χωρίς συμπόνια, με έλλειψη σεβασμού γινόμαστε διπλά θύματα. Απ' τη μία των προβλημάτων μας και απ' την άλλη των σκληρών οικονομικών πολιτικών μπροστά στις ζωές μας. Είναι ζήτημα πολιτισμού των κοινωνιών μας ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με δυσκολίες. Δεν είναι πολιτισμένο να μας αντιμετωπίζουν ως εμπόδιο στην, στην αδυναμία, στην ευκολία και στα κέρδη των εταιριών. Είναι ντροπή ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί έως αυτή τη στιγμή η έκθεση για την πράξη προσβασιμότητα που αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναπηρίας. Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας και τη φωνή μας, να δείξουμε θάρρος και να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας όσο αναλογεί στον κατένα. Μην κρυβόμαστε πίσω από παράλογες πολιτικάντικες και δεν μπορούμε να ξεκαταρίζουμε ούτε τι ισχύει νομικά για το ορισμό των ατόμων με αναπηρία και μην μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στον ορισμό της ομάδας που έχει ανάγκη βοήθειας. Τελευταία η συνάδελφος. Ευχαριστώ. Βεβαίω βρισκόμαστε σε μια έκθεση στα πλαίσια της μεγάλης πολιτικής για την αναπηρία που απασχολεί τα, τον ΟΓΕ εδώ και 25 χρόνια και την Ευρώπη από τη δεκαετία 2000. Η Ευρώπη προτίθεται να αναπτύξει πολιτική για τη μη διάκριση ατόμων με αναπηρία με την ευρεία έννοια ώστε να βελτιώσει και να προωθήσει την ενδοκινητική κινητικότητα. Στους 8 τομείς προτεραιότητας που καθορίζει η δομή του φακέλου έχουμε τρεις δείκτες οι οποίοι είναι συγχυτικοί, δηλαδή δείκτες απασχόλησης, φτώχειας και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν. Και από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αναπτύξει μία μεγάλη σφαιρική πολιτική για την αναπηρία. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μας, ανησυχεί η πρώτη, να μας ανησυχήσει η πρώτη σελίδα της ανακοίνωσης του 2015 που αναφέρει ως γενική ιδέα τη δημιουργία μιας αγοράς που αφορά 120 ε, εκατομμύρια άτομα με πρόληψη το 2010 για, για προσβασιμότητα με 32. Ναι, εντάξει, ε, συμφωνούμε με μια μεγάλη πολιτική για την αναπηρία, όχι όμως την χειραγώγηση, την εμπορική των ατόμων με αναπηρία. που είναι σε μεγαλύτερο μικρότερο βαθμό άτομα τα οποία επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μην πάμε προς ε, μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει η σελίδα 4 της, ε, της έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, θα πρέπει για να δώσουμε από δύο λεπτά μετά ε, να διακόψουμε. Ε, μα, θέλετε αγαπητές συνάδελφοι να ακούσουμε όμως και τους ειδικού. Έχουμε 7 λεπτά για τους τέσσερις ειδικού. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν ήδη. Ήθελα μόνο να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι η έκθεση ισορροπημένη και ρεαλιστική. γιατί μετά από τις συζητήσεις ε, με τους ειδικού. βλέπω πως ε, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ε, ιδέες που δεν είναι ίσως υλοποιήσιμες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όταν διαπραγματευόμαστε με το Συμβουλίο. Και λιγότερο από ένα λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ακούμε την ειδικό την Εμμανουέλ Γκράνζ από την Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, να επιθυμίσω ότι η τωρινή στρατηγική γράφτηκε εν συναρτήσει και αντίστοιχα με τη σύμβαση του ΟΓΕ, παρόλο που δεν την είχαμε επικυρώσει, την είχαμε προσυπογράψει. Οπότε η στρατηγική μα λαμβάνει υπόψη αυτή τη σύμβαση του ΟΓΕ. Βεβαίω η νέα στρατηγική θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή τη σύμβαση του ΟΓΕ και νομίζω ότι αναφέρθηκε αυτό στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ώστε να έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο στη διάθεσή μας και για να προσπαθήσω να πάω και πιο γρήγορα από ό,τι μου είπατε, να σας ευχαριστήσω για όλα τα στοιχεία που αναφέρατε και σας διαβεβαιώνω ότι ο στόχος και για την αξιολόγηση της τωρινής στρατηγικής αλλά και για την εκπόνηση της μελλοντικής στρατηγικής θα είναι να συνεργαστούμε στενά με την κοινωνία των πολιτών και με τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους για αυτή την πολιτική. Αποκλείεται να δουλέψει μόνη τη Κομισιόν σε αυτό το ζήτημα για μια παρόμοια θεματική. Ουδέποτε υπήρχε τέτοιο σκοπό και θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τι συμβολέ σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ακολουθεί η Μακουλάτα Πλασένσια. Ναι. Όχι λάθος, κάποιο λάθος έγινε. Νάτια Χαντάτ. Okay. Thank you. So, um, ναι, Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και πράγματι αν θέλουμε μια ισχυρή στρατηγική και ευθυγραμμισμένη με το ECRPD θα πρέπει να έχουμε τη νέα νομοθεσία η δέσμευση της Ένωσης να είναι ευθυγραμμισμένη με το ECRPD. Μιλάμε για αναπηρία, μιλάμε για προσβασιμότητα. Θα πρέπει λοιπόν στην ε, προσβασιμότητα να μην αποκλείουμε ας πούμε, θέματα όπως η ελευθερία ε, κυκλοφορίας ή μετακίνησης, να μην ξέρουμε τα ακτήρια. Θέλουμε να αναγνωρίζεται παντού αυτό το θέμα της, κινητικότητα και η ελευθερία της ε, μετακίνησης να είναι κάτι το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη σοβαρά. Αλλιώς θα έχουμε βεβαίω μια νομοθεσία χωρίς πραγματική γνήσια προσβασιμότητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα ίδια δικαιώματα για αυτού του ανθρώπους όπως και για όλους τους Ευρωπαίου πολίτες. Οπότε θα πρέπει να επιμένουμε για αυτά τα θέματα προσβασιμότητα και θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε όλα τα άρθρα του CRPD από το 1 μέχρι το 32 για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ροζίτα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Μάριαν Χαρκίν. Δύο πράγματα θα έλεγα για το, ε, που υπάρχουν και να Το ένα είναι στις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της Σύμβασης, όπου έχει ε, δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο κατάλογο του τι θεωρεί ότι λείπει και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να δούμε ακριβώς αυτές τις ε, συστάσεις και να συμμορφωνόμαστε όχι μόνο με το γράμμα αλλά και με το πνεύμα και το δεύτερο που θα έλεγα είναι να δούμε το τι έχουν πει τα μέλη του πλαισίου εφαρμογής. Γιατί αναφέρθηκε ότι είναι σημαντικό να έχουμε σοβαρή παρακολούθηση. Υπάρχει το πλαίσιο και έχει εκφράσει λεπτομερώς πώς την Κομισιόν το τι πρέπει να γίνει. Αυτούς τους δύο τομείς ε, θα έλεγα εγώ ότι χρειαζόμαστε εκεί να εστιάσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι επαφή με το Βελιγράδι. Με ακούτε κύριε Ταντίτς. Ωραία. Δύο λεπτά. Ελπίζω να με ακούτε. Κοιτάξτε. Για την ε, προσβασιμότητα υπάρχει ακριβώς το σχετικό άρθρο που καλύπτει τα περί προσβασιμότητας και καλύπτει το δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες που είναι ανοιχτές στο κοινό. Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει συμμόρφωση με την Σύμβαση των Δικαιωμάτων με Αναπηρία. Λοιπόν, ναι, οι παρατηρήσεις μας είναι ε, ακριβές. Αυτός μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου η κυρία Βουλευτής ε, και να της δώσω και γραπτές απαντήσεις. Λοιπόν, ε, οι παρατηρήσεις είναι αυτές και λένε ξεκάθαρα με ποιον τρόπο πρέπει να κάνει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Και βεβαίως ελπίζω όταν θα εγκριθεί η στρατηγική μετά το 2020. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της ε, συζήτησης. Ε, ευχαριστώ τους ειδικού για τη συμμετοχή. Θα συνεχιστεί η συζήτηση. Το σχέδιο της έκθεσης ε, θα συζητηθεί 30 και 31 Αυγούστου. Η καταληκτική προθεσμία είναι η 6 Σεπτεμβρίου και οπωσδήποτε 28 Σεπτεμβρίου θα δούμε τις τροπολογίες και 19 Οκτωβρίου θα τις ψηφίσουμε στην Επιτροπή για να πάμε στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν μπροστά μας. Και άρα τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και περνάμε άρα στο επόμενο θέμα. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2018. Όλα τα τμήματα. Τον λόγο έχει η εισηγήτρια Ντίρντρι Κλούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουμε πάνω στο σχέδιο και τις γραμμές που γραμμε τον Ιούνιο. Έχουμε εδώ τις προτεραιότητες της ΕΜΠΛ εν ώψη διαπραγματεύσεων. Οπότε, μετά από την δημοσίευση του σχεδίου προπολογισμού για το 2018, και εν αναμονή τη δημοσίευση τη θέση του Συμβουλίου αργότερα σήμερα. Ε, να σου πω ότι το 2018 θα είναι πολύ σημαντικό για την Ένωση, καθώ φτάνουμε στο τέλο αυτή τη εντολή και θέλουμε να αφήσουμε κάτι πίσω μα. Ο προβολισμό είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα και θέλουμε να εξασφαλίσουμε επενδύσει για απασχόληση, για θέσει εργασία. Οι πολιτικές ομάδες ως σήμερα λίγο πολύ συμφωνούν και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις καθώς θα οριστικοποιήσουμε την γνωμοδότηση ε, μέχρι τις 30 Αυγούστου. Συνεχίζουμε να τονίζουμε τα θέματα της ανεργίας των νέων που αντιμετωπίζουν ε, ακόμη και σήμερα πολύ σημαντικά προβλήματα. Φτάσαμε το 2013 στο 24% περίπου, αλλά και σήμερα η ενέργεια των νέων παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σε ορισμένες χώρε ακόμη μάλιστα περισσότερο, αλλά η σύγκριση πάνω και κάτω από το 25 είναι συντηρητικά εις βάρος των νέων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές επίσης μεταξύ κρατών μελών. Ο προβολισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι κάτι θα κάνουμε για αυτές τις μεγάλες διαφορές. Θα καταθέσω και εγώ μερικές τροπολογίες για ομάδες που είναι σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Από εκεί και πέρα έχουμε 73 εκατομμύρια για το πρόγραμμα αλληλεγγύης για τους νέους. Αυτό είναι καλό. Επίσης θέλω να βεβαιωθώ ότι θα προστατευθούν οι γραμμές του προπολογισμού για θέματα απασχόλησης υπέρ όλων των πολιτών και περιμένω, όπως ε, προείπα, σήμερα το απόγευμα τη θέση του Συμβουλίου και ελπίζω ότι θα προστατεύσουν, θα προστατεύσει το Συμβούλιο δηλαδή την πρωτοβουλία για την ενέργεια των νέων. 17 Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Περιμένω τις συνεισφορές σας. Οπότε προς το παρόν σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους συνεισηγητές, τους και συγητές για τη συνεισφορά τους. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά. καθώς και εν ώψη της ψυχορίας στην Επιτροπή μας 30 Οκτωβρίου. Αυτά ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σέτζο Γκουτιέρες για τους σοσιαλιστές. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι που προεδρεύετε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεργαστούμε τόσο ρευστά και ικανοποιητικά όσο στο παρελθόν. Πέρα από κάποιες πολιτικές σκέψεις που ήδη υποβάλαμε για τον προπολογισμό του 18, να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που μας απασχολούν εμάς τους σοσιαλιστές για τον προπολογισμό για φέτος. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνουμε πως οι νέε αναλήψεις υποχρεώσεων και οι νέε πολιτικές και προκλήσεις της Κομισιόν, ιδιαίτερα για θέματα ασφάλειας, άμυνας κτλ. Επειδή αναφέρεται και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, κατά το οποίο μας χαροποιεί, πώς αυτά λοιπόν θα χρηματοδοτηθούν και στο πλαίσιο ποιων προγραμμάτων. Εις βάρος, ας πούμε, του Κοινωνικού Ταμείου θα χρηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πιο ανυποχώρητοι όταν ζητάμε τα νέα εργαλεία αυτά, ώστε να χρηματοδοτούνται με νέα εργαλεία, με νέους πόρους και όχι εις βάρος ανάληψης υποχρεώσεων για προγράμματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, όπως το κοινωνικό ταμείο. Δεν πρέπει λοιπόν αυτά τα νέα προγράμματα, αυτά τα νέα χειρήματα να είναι βάρος κάποιων άλλων. Και δεν χρειάζεται να πούμε ποιο χρειάζεται περισσότερο και ποιο λιγότερο. Όλα είναι εξίσου απαραίτητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή ιεραρχήσεις. Επίσης για τον προπολογισμό για του χρόνου Έχουμε μείωση στο ΤΕΒΑ όσον αφορά στην αλήψη υποχρεώσεων στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Αυτό σε μια στιγμή βέβαια που αρχίζουμε να βγαίνουμε σιγά σιγά από την οικονομική κρίση και φαίνεται ότι είναι λιγότερο σημαντικό το να κάνουμε κάποιες ε, προσπάθειες στα πλαίσια αυτών των ταμείων όπως το ΤΕΒΑ. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενισχύσουμε το ΤΕΒΑ γιατί η ύφεση συνεχίζει να υπάρχει στο περιθώριο των κοινωνιών μας και αφορά ανθρώπους που χρειάζονται τα απαραίτητα, δηλαδή τροφή και ένδυση για να ζήσουν με κάποια ελάχιστη αξιοπρέπεια. Οπότε θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτή τη μείωση του 9% στο ΤΕΒΑ. Επίσης, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας για την Παγκοσμιοποίηση θεωρούμε ότι και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί, αντί να υποχωρήσει. Και κατά λίγο, Πρόεδρε, όπως ξεκίνησα λέγοντας, ότι είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τρόπο ρευστό με την εισηγήτρια και τους προσώπους των υπολείπων πολιτικών ομάδων, όμως είναι απαραίτητο εμείς στην Επιτροπή αυτή να προσπιστούμε σημαντικά εργαλεία όπως το ΤΕΒΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, δεν βλέπω την Ουλρίκη Τρεμπέζιους. Λοιπόν, Μάριαν Χάκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή. Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά ως τώρα. Χαίρομαι διότι η εισηγητρία στην έκθεσή της, στη γνωμοδότηση, μάλλον έλαβε υπόψη της στα σχόλια της Επιτροπής. Βλέπω μια προσπάθεια προστασίας των γραμμών για την απασχόληση. Ε, με αφορμή αυτό που είπε και ο Σέτζιο είπε για τη χρηματοδότηση του σώματο Αλληλεγγύης το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορα εφιστεμένα πράγματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τη συλλογιστική. Εδώ βλέπουμε περικοπές στο κοινωνικό ταμείο, στο πέρασμος. Υπάρχει πιο νούμερο. Τι, τι περικόπτεται και πού. έχουμε κάποια εκτίμηση ότι τα κονδυλία που περικόπτονται θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα κάπου αλλού. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά. Επειδή κάποιο μα είπε ότι αυτή η ιδέα τη ελληνική είναι καλύτερη, δεν λέω όχι, αλλά πού πηγαίνουμε, χωρί χρηματοδότηση, χωρί νούμερα, πού θα βρεθούν τα χρήματα, από πού θα περικοπούν. Και στην παράγραφο 7 συγκεκριμένα τώρα, Η ζωηρθογραφή είναι λίγο αμφίβολη. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω όλα αυτά γιατί βλέπω περικοπές στο πρόβλημα. FEED. Ε, υπάρχει κάποια ανάλυση. Πού βασίζονται όλα αυτά. Δηλαδή πώς τεκμηριώνονται και πώς δικαιολογούνται αυτές οι περικοπές, ότι θα έχουμε περισσότερη προστιθεμένη αξία αν τα χρήματα αυτά πάνε αλλού. Δεν θα δώσω αναγκαστικά τώρα μάχη γι' αυτό, αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω πράγματα να αποφασίζονται, να προτείνονται χωρίς, να, ε, χωρίς εξήγηση, χωρίς να ξέρουμε γιατί κάνουμε τι. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον Ζωάο Λόπες, δεν βλέπω την Τζιν Λάμπερτ το FDD δεν όρισε κάποιον, οπότε έχουμε τον Ντομινίκ Μαρτάν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν εκπλήξεις εδώ τώρα, εν ώψη 18. Δυστυχώ διαπιστώνουμε τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Περισσότερη ενεργεία, περισσότεροι νέοι άνεργοι, οι μικρομεσαίες είναι σε χειρότερη κατάσταση, κλείνουν, οι όλο και περισσότεροι μετανάστες, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, περισσότερη φτώχεια και το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται με φτώχεια και αποκλεισμό, με κοινωνικό αποκλεισμό, είναι σε εκρηκτικά επίπεδα. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τα αίτια, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα με ασπιρίνες. Το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Ευρωπαίους σε ακραία ένδια κλπ. Αυτά και, και τώρα ξαφνικά ειδική, ο δικός μηχανισμός για τους νέους. Αυτά νομίζω ότι είναι αναποτελεσματικά και καταδικασμένα σε αποτυχία. Οι διαπιστώσεις, επαναλαμβάνω, είναι οι ίδιες. Διαβάστε από προπολογισμό σε προπολογισμό, δεν αλλάζει τίποτα. Μήπως ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε. Και ένα άλλο ερώτημα είναι πώς θα αντισταθμιστεί η, η απώλεια της Βρετανικής συνεισφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην Κομισιόν. Καλωσορίζω την Μπριγκίτε Φελάχη και την Πανασκαλίνη Βέρεχε. Φιλ... φυλάχη, Φιλάχη βλέπω εγώ ότι θα μιλήσει. Δεν ξέρω. Απαντήστε βεβαίως και στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. τη λέγομαι. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για το σχέδιο γνωμοδότησης που, όπως πάντα θα έλεγα, θέτει τα σωστά ερωτήματα σχετικά με το σχέδιο προπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τα, τις προτεραιότητες του προπολισμού. Να απαντήσω αυτής αμέσως σε ερωτήματα που έθεσε η συγκήτρια και οι ισχυώδεις συγκητές. Το σχέδιο προπολισμού της Κομισιόν επιβλήθη κατόπιν λεπτομερούς και σε βάθος αναλύσεως των θεμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εκεί ζητούμε κονδύλια, τα οποία θεωρούμε στον προπλησμό ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Η μείωση κάποιων κονδυλίων δεν πρέπει να ενισχύει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Τόσο λοιπόν στο Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση όσο και αυτό για τους Ευρωπαίους ακραία ε, δεν υπάρχει ανησυχία. Όσον αφορά το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Είναι μια νέα πρωτοβουλία, η οποία όπως σε όλες τις περιπτώσεις νέων πρωτοβουλίων ε, γύρει βεβαίως ερωτήματα. Είναι πρωτοβουλία πάντως που πολιτικός είναι σημαντική, διότι είναι, αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια μικτού χαρακτήρα πρωτοβουλία, με την έννοια ότι συμμετέχουν και εθελοντές αλλά και συνεπάγεται τοποθετήσει νέων σε επιχειρήσεις οι οποίοι εκεί βρίσκουν απασχόληση ε, στο πλαίσιο μαθητείας. Θα λέω ότι πρόκειται για συνδυασμό προγραμμάτων και ξέρετε, όπως με όλες τις νέες ε, πρωτοβουλίες έχουμε και 25% νέα κονδύλια μέσα από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Λοιπόν, πρόκειται για νέα πρωτοβουλία, η οποία χρηματοδοτείται και ε, με νέο χρήμα, αλλά και με μεταφορά κονδυλίων από άλλε γραμμέ. Εδώ αξιοποιήσαμε προγράμματα που ήταν λογικό να χρησιμοποιήσουμε. Ήταν οι φυσικές, αν θέλετε, πηγές. Το Erasmus Plus, το οποίο είναι συναφές. Άρα λοιπόν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των δύο προγραμμάτων και όσον αφορά την απασχόληση και την τοποθέτηση νέων εργαζομένων αυτό γίνεται μέσω και των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου συνοχή, 35 εκατομμύρια εκεί για μια τριετία από το Κοινωνικό Ταμείο μικρή συνεισφορά αλλά είναι σημαντικό πιστεύω και το Κοινωνικό Ταμείο να συνεισφέρει εδώ γύρω στα τέλη του πολιτούς πλαισίου. Οι στόχοι τώρα. Νομίζω ότι έχουν εκλογικευθεί. Προκρίνουμε την ένταξη στον τομέα της απασχόλησης, ένταξη στην αγορά εργασίας αυτών των νέων και ελπίζουμε, ελπίζουμε ότι η βασική πράξη θα εγκριθεί από την Κομισιόν και θα προβληθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι μια νομοθετική προτεραιότητα για φέτος. Η νέα αυτή πρωτοβουλία πάντως για τους νέους ελπίζω ότι και αυτή θα πετύχει γιατί το αξίζει. Αυτά ελπίζω να κάλυψε τις περισσότερες, να απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε μια διόρθωση. 14 Ιουλίου τροπολογίες με email ε, για τις ε, τροπολογίες για το σχέδιο έκθεσης 17 Ιουλίου. Προφανώς είναι ένα θέμα software. Γι' αυτό απαιτείται περισσότερος χρόνος. Ελπίζω λοιπόν να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα. και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε κανονικά. Αυτά. Οι συντονιστές θα μιλήσουν πέμπτη απόγευμα με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε και νωρίτερα. Καλό διάλειμμα εύχομαι. Τρεις η ώρα ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Έχουμε λίγη δουλίτσα. Ελπίζω να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Καλή όρεξη.